Συνάδελφοι, θα πρέπει να είμαι, να θυσιαστώ σήμερα το πρωί και γι' αυτό θα ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες ως το δυνατόν συντομότερα. Έχουμε πολλές, οπότε θα ξεκινήσουμε αμέσως. Παρακαλώ να κάνετε τη δοκιμή, να κάνουμε τη δοκιμή της κάρτες. Είμαστε έτοιμοι. Right. Uh, the first is the report progress. Πρώτα απ' όλα θα ψηφίσουμε. Όχι, θα πάρει πολλή ώρα να πάτε και να ξανάρθετε. Όταν ε, ξεκινάει κανείς μια επιχείρηση πρέπει να έχει και μια λύση, μια στρατηγική για την διέξοδο, τη λύση. Έτοιμη. Έχουμε ακόμα τρει-τέσσερι συναδέλφου που υπογράφουν. Βιαστείτε παρακαλώ γιατί θα αρχίσουν οι ψηφοφορίε. Please hurry up. Βιαστείτε. Can sign also. Μπορείτε να υπογράψετε και μετά. Παρακαλώ. Έκθεση προόδου σχετικά με τη Βοσνία Ριζακοβίνη. Ησυχία παρακαλώ. 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ 16 υπέρ Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ας κάνουμε έλεγχο για τη 16. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Okay, those Κάποιοι θέλουν να μας να αποφασίσουν πόσο, πόσο, πόσο θα ψηφίσουν. Okay, so it... Πέρα τη απορρίφθηκε. Εντάξει, καταγράφουμε και τις δικές σας ψήφους. So it's 18. 18. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 17. Υπέρ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 κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ κατά αποχές να το ελέγξουμε. 44 ist das, ne? Die, Antrag, die Abstimmung ist geschlossen. Πέρας ψηφοφορίας. 29 αρνητικές ψήφοι, 19 υπέρ, απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην τροπολογία, την προφορική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 48. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εντάξει, να το ελέγξουμε αν θέλετε. Ελέγχουμε τη 48. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Abstimmung ist geöffnet. Ist Πέρας ψηφοφορίας, 43 ψήφοι υπέρ, 10 ψήφοι κατά. Εγκρίνεται. Ποιος είπε να το ελέγξουμε? Ένα βαθμό μείον θα σας αφαιρέσουμε. Ε, ναι, αλλά θα πρέπει οι μεγάλε ομάδε να σηκώνουν καλύτερα τα χέρια του για να βλέπουμε, πρόεδρε. Λοιπόν, 50 ε, συγγνώμη, υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. 51 υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. 52 υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. 53 υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. 54 υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. 55 υπέρ, κατά, αποχές Να το ελέγξουμε. Τώρα θέλω εγώ να το ελέγξουμε. Την 55 ψηφίζουμε. Ja. 26 υπέρ, 30 κατά. Ποιο ήτανε, ποια, ποια ψηφίσαμε? Την 55. Λοιπόν, συμβαστική 5 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 69. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 70. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 71. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 72. Χωριστή ψηφοφορία. Για το πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στην 73. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 74. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 75. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 76. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 77. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 78 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 79 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 80 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 82 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 84 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 85 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία της ε, εισηγήτριας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 88 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται προφορική τροπολογία 4 υπέρ, 4, 4, 4, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 92, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 93, υπέρ. Α, να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 92 ηλεκτρονικά. Again. The Greens? Is closed. It's closed. 25 ψήφοι υπέρ, 31 κατά, απορρίπτεται. 93 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 94 υπέρ, όχι, όχι, συγγνώμη, 97 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 98 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 98 υπέρ, κατά. Την 98 την κάναμε. 99 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε στην παράγραφο 28α, τροπολογία 100, υπέρ, κατά, εγκρίνεται, συγχαρητήρια. 101, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2, υπέρ, κατά, αποχές, ξανά. Ποιος είναι υπέρ της 2, 2, υπέρ, κατά, Ποιο εγκρίνεται, αλλά να το ελέγξουμε. Εγκρίνεται, αλλά α ψηφίσουμε ηλεκτρονικά τη 2. Ε, ναι. äh, Πέρας ψηφοφορία. 32 ψήφοι υπέρ, 30 κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται.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 την ε, έκθεση. Πέρα Abstimmung Πέρας ψηφοφορίας. «58 ψήφοι υπέρ και 2 ψήφοι κατά». Θα τους βρει τους δύο οι Ντόρες, είμαι σίγουρη. Είμαι σίγουρος.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 Λοιπόν, τώρα θα έχουμε τη διασκέδαση να ψηφίσουμε την έκθεση της κυρίας Όμεν Ράιτεν. Νομίζω ότι είναι λίγο περίπλοκα τα πράγματα και προσέξτε παρακαλώ να σηκώνετε τα χέρια σας για να αποφύγουμε πολλές ηλεκτρονικές ψηφοφορίες. Να γνωρίζουμε δηλαδή διανατάσεως της χειρός περίπου που είναι τα πράγματα, να μην αναγκαζόμαστε κάθε φορά να κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Κύριε Όμεν, θέλει το λόγο για μια παρατήρηση. Ντόρις, ποτέ δεν με κατάλαβες τώρα. Σήμερα θα με καταλάβεις. Ο κύριος Ομπιόλς, εξ ονόματος της ομάδας μας κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να προτείνω μία προσθήκη στη συμβιβαστική τροπολογία υπαριθμών 20 στην αρχή θα παρακαλούσαμε να προσθεθούν οι λέξεις εντός εισαγωγικών σύμφωνα με τις αρχές του διεθνούς δικαίου. In accordance with the principles of international law. Και νομίζω ότι θα συμφωνήσει και η Δεν φαντάζομαι να διαφωνεί με την πρόταση αυτή. Yeah. Ναι. Η κυρία Φλότρου, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να προτείνω στην εισηγήτρια για την Συμβαστική 18 ότι είμαστε διατεθειμένοι να υπερψηφίσουμε αρκεί να διευκρινιστεί ότι η σύμβαση για το ναυτικό δίκαιο είναι μέρος του κοινοτικού δικτυού. Δεν είναι μέρος είναι μέρος του κοινοτικού κεκτημένου. Εν μέρη αποτελεί μέρος του κοινοτικού κεκτημένου. Yeah, Κύριε Όμεν, σε αυτό το κείμενο, εγώ προτιμώ το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν δέχομαι αυτή την προφορική τροπολογία για το δίκαιο της θάλασσας. Δηλαδή, είναι σήμα ποιότητα τώρα η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ωραία, τότε θα το ψηφίσουμε, όχι συμβαστικά. Ε, συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 74, wer ist dafür? 74 υπέρ. Κατά. αποχέ, απορρίπτεται. 76 υπέρ. Κατά. Αποχέ απορρίπτεται. 78 υπέρ. Κατά. άποχε, απορρίπτεται. 79 υπέρ. Κατά. άποχε, απορρίπτεται. 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Η 82 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 83 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Και τώρα θα έρθουμε στην 87 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 89 σε τρία τμήματα. Τμήμα πρώτον υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τμήμα δεύτερο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τμήμα τρίτον υπέρ κατά Εδώ χρειάζεται έλεγχος τώρα. Are you in favor? What are you, what is your position? In favor. In favor. Okay. Was ist das? Die Abstimmung ist geschlossen. Απορρίπτεται. 27 υπέρ, 35 κατά. 91. 91 τμήμα πρώτον. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απόρριψετε. Τμήμα δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 92 τμήμα πρώτον υπέρ. Κατά. Αποχές. απορρίψετε. Τμήμα δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές. απορρίψετε. Η συμβιβαστική 3. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ερχόμαστε λοιπόν στην 97 υπέρ. Κατά αποχές απορρίψετε. 99 υπέρ. Κατά αποχές απορρίψετε. 101 πίπτη. έτσι κι αλλιώς Οπότε ερχόμαστε στην 104 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 106 υπέρ. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 110 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η συμβαστική 4 υπέρ. Dagegen Κατά αποχές εγκρίνεται. 116 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 120 σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές. Νομίζω ότι έχει εγκριθεί. Θέλετε έλεγχο. Παρακαλώ. Σλούς. 37 υπέρ, 28 κατά, εγκρίνεται. 121 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 122 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 123 υπέρ. Κατά αποχές απορρίψετε. Η συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 138 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 141 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι έχει εγκριθεί αλλά μάλλον χρειάζεται έλεγχο γι' αυτό Όντως, 36 υπέρ, 30 κατά συμβαστική, 8 κατά πίπτη, επειδή εγκρίθηκε η συμβαστική 7. Όχι, την ψηφίζουμε. Η συμβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 144 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έλεγχο. Ας την ελέγξουμε λοιπόν. Πέρα.

Το πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα τι έχουμε, 149, όχι, 154 πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, άποχες εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα υπέρ, Α, όχι, έχει διεκπαιρεθεί μάλλον. Η συμβαστική 9. Α, όλα έχουν εγκριθεί. Μάλιστα. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η συμβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 155 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η συμβαστική 9α Κατά αποχές εγκρίνεται. 174. Το δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και ερχόμαστε στις τέσσερις τροπολογίες όπου τέσσερις άνθρωποι είχαν την ίδια σκέψη ακριβώς. Μάλλον έχουν όλοι τον ίδιο συνεργάτη. Ο πρέσβης δεν ήταν. Ψήφι υπέρ αυτής της συλλογικής τροπολογίας, υπέρ κατά άποχες. Δηλαδή μόνο οι συντάκτες βασικά.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 189 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 190 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 191 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 192 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η συμβαστική 10 τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία παρελθόν 200 επέ. κατά αποχές απορρίπτεται. 201 επέ. κατά αποχές απορρίπτεται. 122 εγκρίθηκε, δεν θυμάμαι. Ωραία. Ψηφίζουμε 203 υπέρ. Σε δύο τμήματα μάλιστα. Τμήμα πρώτον. Υπέρ. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα της 203 υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. Και το τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Από... Εγκρίνεται πίσω. Η συμβαστική 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η συμβαστική 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η τροπολογία 214 τώρα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η συμβαστική 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2.19 υπέρ κατά αποχές νομίζω είναι σαφές. Θα ψηφίζουμε τη 2.19. Υπέρ κατά... Οι φιλελεύθεροι δεν ψηφίζουν, τι γίνεται. Έλεγχο θέλετε, καλά. Ας επαληθεύσουμε. Για να πιο εύκολη ζωή του κυρίου Λάμστορφ, όχι τίποτα άλλο. Πέρας. Απόρριπτεται 22 υπέρ 43 κατά. Και τώρα, πού πάμε. 220 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 222 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 225 τμήμα πρώτον υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Το δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 228 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 229 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 213α ε, συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 233 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 234 ε, ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 235 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 238 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 240 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 242 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και τώρα ερχόμαστε στη συμβιβαστική 14 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 247 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ερχόμαστε στη 254 κύριε Λάτφορτ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 257 τμήμα πρώτον υπέρ κατά κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ...258 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 261 Κατά τμήματα, τμήμα πρώτο υπέρ, κατά, ξανά. Δύο τμήμα πρώτον υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 16 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 264 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 266 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 267 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 269 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ερχόμαστε στη 275 υπέρ κατά ξανά παρακαλώ 275 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 277 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 278. 277 τι γίνεται. Θέλετε έλεγχο, ορίστε. Επαληθεύουμε τη 277. Οι πράσινοι χάνουν δύο πόντους. Πέρας. Ναι, ήταν ε, μικρή διαφορά, δεν φαινόταν. 2,78 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίθηκε. Είχε εγκριθεί το κύριος. Ε, τουλάχιστον όσοι ψήφισαν. 2,80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 281 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 282 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 283 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 284 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 285 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 286 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 287 ε, υπέρ κατά εγκρίνεται äh, Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 36 προς 22. Πάμε στην 289. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 290. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 281. Υπέρ. 291. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 294 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 295. Την 92 την εγκρίναμε. Ναι, έχουν συγχωνευτεί, αλλά την ψηφίζουμε. 2,95 λοιπόν, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 18, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 297 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 298 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 298 υπέρ κατά όχι. Α, όχι. 2,99. 2,99. Ποιος είναι υπέρ της 2,99. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 300 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 301 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 302 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 303 υπέρ. Κατά. Οι σοσιαλιστές απορρίπτεται. 304 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 305 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 306 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 307 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 308 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 309 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 310 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 311 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 312 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 313 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 314 και 315 υπέρ Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 3.16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. πρέπει να την ψηφίσουμε τώρα αυτή, έτσι. Ναι. Λοιπόν, μόνο για, τους, για τον όρο in parallel θα ψηφίσουμε. Ποιος είναι υπέρ. κατά, αποχές, να το ελέγξουμε, αλλά μάλλον εγκρίνεται. Παρόλο που πολύ λυπάμαι. Original, paragraph 23. Παράγραφος 23, original. Πέρας ψηφοφορίας. Εντάξει, εγώ ψήφισα λάθος, αλλά δεν αλλάζει και τίποτα. Α, τελικά σωστά είχα ψηφίσει. Όχι, όχι, λάθος, λάθος ψήφισα, αλλά δεν αλλάζει τίποτα. Στην ουσία τη υπόθεση. απορρίπτεται. Ψήφισα λάθος, αλλά το αποτέλεσμα βγήκε σωστό τελικά. 3.17. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3, 17 ε, δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3.18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3.19. Υπέρ. Κατά. αποχέ. Νομίζω εγκρίνεται. Το ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Mm? ist geschlossen. Πέρασε ο φορέα. Απορρίπτεται 26 προς 39. Falls 294 angenommen. Τη 294 η 321 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στην 3.36. Υπέρ. 3.37. Ναι, αλλά εδώ λέει 3.36. Λάθος είναι ο κατάλογος. Ωραία. Πάμε στο 3.37. Άρα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3.42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3.43 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3.44 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3.45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 346 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 347 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 348 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 349 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 350 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 351 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 353 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 355 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Να το ελέγξουμε. Παρακαλώ το ΕΛΚ να συμμετέχει στην ψηφοφορία. Η Abstimmung ist geschlossen. Πέρας ψηφοφορία. 3.55. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται 29 προς 32. Πάμε στην 356 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 359 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 363 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 363. Απορρίπτεται σαφέστατα. Αν επιμείνεις θα βγουν τρεις πόντοι από τη βαθμολογία σας. Λοιπόν, 364, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τρία, εξήντα θέλετε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 364. 18 προ 49. Απορρίπτεται. 3.65 λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3.66 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3.67 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 368 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 369 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 370 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 371 υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε. Schließen. Πέρας. 23.43. Απορρίπτεται. 3.71 ψηφίσαμε, έτσι. Ωραία. 3.72. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3.73. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3.74. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 3.75 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 3.76 3.76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 3.78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 3.79 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 380 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 381 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβεβαστική 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 387 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. 389 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Μετά πάμε στην 398. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 399 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 409 υπέρ κατά αποχές Ε, δεν μπορούμε τώρα να το κάνουμε αυτό στον κύριο Κασουλίδη. Απορρίπτεται. Πάμε στην 411. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4.13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 4.14-4.15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές.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 αποχές απορρίπτεται. 19 υπέρ κατά να το ελέγξουμε. Υπέρ της 19 κατά απορρίπτεται. 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 25 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 30 υπέρ. Α, ε, καταπίπτει. Α, 31 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 32 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 33 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 34 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 35 υπέρ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 αποχές απορρίπτεται. 47 υπέρ κατά αποχές δεν ήταν σαφές. 47 πάλι, σηκώστε τα χέρια σας, υπέρ. Α, α, άντε να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Περίπου έκλεισε η ψηφοφορία, τώρα έκλεισε. Απορρίπτεται. 49. 48, συγγνώμη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 49. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 50. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται.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 αποχές απορρίπτεται. 63 με την αλλαγή υπέρ 36, 63 ε, συγγνώμη, 63 ε, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 65 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 66 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 67 υπέρ, κατά, αποχές Απορρίπτεται. Και τώρα πάμε στην ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σύνολο της έκθεσης. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η έκθεση 54 ψήφι προς 4. αλλά δύο παραπάνω αρνητικές ψήφοι από αυτή της Ντόρης. Κυρία Όμεν, θα ήθελα να ευχαριστήσω όχι μόνο τους σκιώδης ηγητές, αλλά και τους συνεργάτες και βοηθούς τους και το Γιουρούν, το Γιάνν Βίλεμ και το Λούκα Τιπέτρο γιατί ήταν πάρα πολύ σκληρές οι διαπραγματεύσεις, χρειάστηκαν πάρα πολύ χρόνο, αλλά καταλήξαμε σε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα και σας ευχαριστώ. Hmm? Sir Robert. Sir Robert. Atkins. Sir Robert Atkins. Πρόεδρε, ένα μικρό διαδικαστικό. Ποιο ακριβώς είναι το καθεστώς μιας τροπολογίας που προτείνεται από, το από τον Υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου όταν δεν είναι πλέον μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, είναι τιμητική λεγόμενη τροπολογία. Exactly. For the entire career. Wir kommen damit jetzt zu dem Bericht Brandner. Ερχόμαστε στην έκθεση Echt Έχετε να πείτε ένα τελευταίο λόγο πριν σοπάσετε για πάντα. Das ist nicht der Fall. Wir... Όχι. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα στην απόφαση του δικαστηρίου. Ε, η τροπολογία 1 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 73 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Σα παρακαλώ ησυχία εκεί πίσω στι ορεινέ φθηνέ θέσει τη αιθούση. Η συμβαστική 1 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. ερχόμαστε στην 94. Ψηφί Κατά αποχές εγκρίνεται. 96 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 97. Τμήμα πρώτο υπέ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 98 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Από το ΕΛΚ ψήφισαν μόνο δύο. Δεν βλέπω χέρια. 99 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 100. Το πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 101 υπέρ. Απόφαση. Κατά αποχές εγκρίνεται. 102 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Όχι λέει η κυρία Μπράντνα. Ως είπατε. 102. Δεν εγκρίθηκε. Ας το ελέγξουμε τότε. Πέρας ψηφοφορία Απορρίπτεται 16 υπέρ 28 κατά. Πού είχαμε μείνει. Συμβαστική 3. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 107. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 108 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 109 υπέρ. Οι σοσιαλιστές σηκώνουν χέρια στο όχι. Αν είναι αργή εγώ τι φταίω. 109. Υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. 110 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίψτε 111 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 112 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 113 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η προφορική υπαρχόν 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 114 υπέρ. Συγγνώμη, διορθώνει ο Πρόεδρος. 115 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 12 της ανάπτυξης υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 5. Κατά λέει ο Πρόεδρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται εγκρίνεται ρήμην του ΕΛΚ που δεν ψηφίζει. Μόνο συνάδελφος Πέτερινγκ από το ΕΛΚ ολόκληρο ε, ψήφισε και ουδής άλλος. του το μετράμε θετικά αυτό, του πιστώνεται. 119 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έχουμε τη δέκα τώρα της Επιτροπής Ανάπτυξης, με τα 2, τμήμα πρώτον υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τώρα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η προφορική υπαριθμών 4 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 123 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 124 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 125 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 129 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 130 υπέρ. Απερίφθη, διότι αυτή τη φορά οι φιλελεύθεροι την καταψήφισαν. 130 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 131 Είπε. κατά αποχές εγκρίνεται. Η 130 εγκρίθηκε είπαμε, άρα καταπίπτει η επόμενη. δε DV11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 133. Δύο τμήματα, τμήμα πρώτο Είπε. κατά αποχές απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 134 υπέρ. Κύριε Πόσελτ, μην αποσπάτε από τα καθήκοντά του τον κύριο Πέτερινγκ. 135 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 135 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 136 υπέρ κατά η συγγήτρια ζητεί το λόγο 136 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Μπέρντ Πόσελτ σε παρακαλώ πραγματικά ενοχλείς τώρα που είμαστε 136 η κυρία Μπραντνερ ε, σας ευχαριστώ θα ήθελα να κάνω μια προφορική τροπολογία εδώ. Το τρίμηνο να γίνει εξάμηνο. Οι τρεις μήνες έξι. 137. Σε έξι μήνες τότε όμως. Η ψηφιπέ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ερχόμαστε στην τροπολογία 35 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 36 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. προφορική 6 υπέρ. Κατά απορρίπτεται. ΔΕΒΕ 3 υπέρ κατά άποχες δεν είναι σαφές τουλάχιστον εγώ δεν το κατάλαβα η ε, τρία της Επιτροπής Ανάπτυξης Η Abstimmung ist Πέρασε. Απορρίπτεται 14.30. 37 είπε, Κατά αποχές απορρίπτεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθεται. 39 τώρα την ψηφίσαμε. ΔΕΒΕ 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η προφορική 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σαν τα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική 9 υπέρ. Κατά. Κατά. Εγκρίνεται. Και τώρα. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η προφορική 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Απορρίπτεται, συγγνώμη. 9 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. ΔΕΒΕ6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. ΔΕΒΕ7 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. ΔΕΒΕ8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχο θέλετε. Ψηφίσατε. Ψηφίζουμε τη συμβαστική παριθμόν 10. Πέρας. 30 υπέρ, 17 κατά εγκρίνεται. 62 υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. 63 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 64 ειπε κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 70 υπέρ κατά αποχές Δεύε DV5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 77 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται.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 κατά αποχές εγκρίνεται. Η 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 12 υπέρ τσεκ. Ας ελέγξουμε την 11 λοιπόν ηλεκτρονικά. Απελευθεύουμε. Ναι, έχετε δίκιο. Εγκρίθηκε. Ε, γιατί βλέπω ότι έχω εκτιμήσει λάθο του σοσιαλιστές, αλλά όλη μου τη ζωή πέφτω έξω με του σοσιαλιστές. Εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Και τώρα έχουμε στην οπολογία 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 19 υπέρ. Τις απολογίες κυρίας Νέντσκι μπορούμε να τις ψηφίσουμε όλες μαζί. Όχι, 19 υπέρ. Κατά άποχες απορρίπτεται.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 ηλεκτρονικά τώρα το σύνολο του έργου τέχνης. geschlossen. Πέρας. Α, εσείς κυρία Μπράντερ, είστε ακόμα χειρότερα από τις υπόλοιπες δύο συναδέλφους. Έχετε πέντε ψήφους κατά. Ε, συγχαρητήρια, εγκρίνεται. Θα πρέπει να συστήσουμε όμως και υποεπιτροπή δικαιώματα των ανδρών να αναλαμβάνουν και καμιά έκθεση καμιά φορά. Ε, European oh, ah. Which are you here in that body or what is it? No, just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 Meine Damen und Herren, Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, έχω τη μεγάλη τιμή να καλωσορίσω εδώ τον δόκτωρα Βέρνερ Χόιερ, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, που θα συζητήσει μαζί μας ε, ιδιαίτερα για θέματα της χρηματοδότησης εξωτερικής πολιτικής. αυτό τον καιρό. Συζητούμε και για τα χρηματοδοτικά μέσα με το Συμβούλιο και είναι πάρα πολύ επίκαιρο να ανταλλάξουμε απόψεις για να συμπεριλάβουμε και τις δικές σας θέσεις και να οργανωθούμε πρακτικά καλύτερα από ό,τι ενδεχομένω είχαμε πράξει στο παρελθόν. Χαίρομαι που στο πρόσωπο του κυρίου Χόε έχουμε κάποιον που διατέλεσε δύο φορές αναπληρωτής υπουργό Εξωτερικών ε, της Γερμανίας και μάλιστα και στην ε, Βουλή, τη Γερμανική, στον Bundestag, ήσασταν στην ε, Επιτροπή Εξωτερικών. Ε, άρα με διπλή ιδιότητα έχετε μελετήσει αυτά τα θέματα. Υπάρχουν προβλήματα και ανισορροπίες όχι μόνο στην Ευρωζώνη αλλά και στην πολιτική γειτονίας και αυτά παίζουν ρόλο. Έχουμε διαφορετική ανάπτυξη κατά τόπους και είναι ενδιαφέρον να ακούσουμε με ποιο τρόπο και τα χρηματοδοτικά μέσα και οι δραστηριότητε τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αλλά και άλλων μπορούν να συνδεθούν ενδεχομένω. για να επιτευχθούν έτσι καλύτερα αποτελέσματα και να μην έχουμε παράλληλες ε, ή αντιφατικές ε, δραστηριότητες. Έχετε το λόγο κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, Αξιότιμες κυρίες και κύριοι βουλευτές, σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια και τη φιλική υποδοχή που με επιφυλάσσετε. Έχουμε ασχοληθεί τα τελευταία 25 χρόνια περίπου από κοινού τα θέματα αυτά που μας απασχολούν και μεγάλη χαρά Είχαμε πάει μαζί και στη Λισαβόνα, λέει εγώ, από ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ε, ε, ο κύριος Χόιερ από τη γερμανική κυβέρνηση για να διαπραγματευτούμε τη συνδίκη της Λισαβόνας. Ωραία. Χαίρομαι λοιπόν που έχω την ευκαιρία να σας παρουσιάσω κάποια θέματα για τα οποία τώρα έχω την αρμοδιότητα και θα πέρασω στα αγγλικά. Εδώ και κάποια χρόνια ο πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει έρθει ξανά και ξανά εδώ για να συζητήσουμε με τον πρόεδρό σα, τον κύριο Μπροκ, και τον ευχαριστώ που μου έδωσε και σήμερα αυτή την ευκαιρία να είμαι κοντά σας. Μαζί με την κυρία Τόμ Μπάρτεν στα αριστερά μου, που είναι Γενική διευθυντή για τι δραστηριότητε εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Μαζί θα διαμορφώσουμε τη νέα εξωτερική εντολή της ε, Ευρωπαϊκής Τράπεζα Επενδύσεων για το 2014-2020. Ελπίζω έτσι να καλύψω και κάποιες απορίες που μπορεί να έχετε σχετικά. Μαζί με τα κράτη-μέλη θα αποφασίζετε εσείς πώς η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα στηρίξει την εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ερχόμενα 7 χρόνια. Εξωτερικές πολιτικές που κάποιοι φοβούνται ότι θα πέσουν θύματα της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης και τη επικέντρωση τη Ευρωπαϊκή Ένωση στα εσωτερικά τη προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, είναι καθοριστικό το διάστημα αυτό για την Ευρώπη και δεν έχουμε χρόνο για να εφησυχάσουμε. Ζούμε σε ένα περιβάλλον όπου τα κέντρα εξουσία συνεχώ αλλάζουν και οι παραδοσιακέ γεωπολιτικέ ε, τάσει δεν ισχύουν πλέον. Η Ευρωζώνη είναι η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου και η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ο μεγαλύτερο εξαγωγό και εισαγωγό ε, εμπορευμάτων. Όμω ε, χάνει το πρωταγωνιστικό τη ρόλο, κυρίω λόγω των αναδυόμενων αγορών και ιδιαίτερω λόγω τη Ασία. Το βασικό ερώτημα είναι, είμαστε έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε τι προκλήσει τη παγκοσμιοποίηση. Η Ευρώπη μπορεί να παραμείνει ένα ελκυστικό προορισμό, ανταγωνιστικό και στην μπροστοφυλακή των τεχνολογικών εξελίξεων. Οι προκλήσει πάνω απ' όλα είναι οικονομικού χαρακτήρα, αλλά οι επιπτώσει είναι και πολιτικέ και ε, συνέπειε ασφαλεία αλλά και πολιτιστικέ. Η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση και από τι δύο πλευρέ του Ατλαντικού έχει οξύνει τον ε, διεθνή ανταγωνισμό. Οι αναδυόμενε αγορέ έχουν μεγαλύτερη οικονομική και γεωπολιτική επιρροή. Η τάση είναι να δημιουργείται ένα κόσμο με πολλού διαφορετικού πόλου και να ε, χάνουν σε αυτόν τον ανταγωνισμό η Ευρώπη και οι Ηνωμένε Πολιτείε που τον έχουν αρχικά επιταχύνει. Οι αναδυόμενε χώρε και ιδίω οι πιο πολυπληθεί όπω η Κίνα, η Ινδία, η Βραζιλία έχουν αυξήσει το βάρο του ε, ε, στο διεθνή σχεδιασμό πολιτική. Σήμερα οι συναντήσει του G20 είναι πιο σημαντικέ από του G8. Το ΑΕΠ τη Κίνα για πρώτη φορά έχει ξεπεράσει τα 8-3 δολάρια. Είναι το 55% του ΑΕΠ των Ηνωμένων Πολιτειών. Και η οικονομία τη Κίνα προβλέπεται να αυξηθεί κατά 8% φέτο. Και πάλι, αυτή είναι η γεωπολιτική πραγματικότητα σήμερα. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι η Ευρώπη θα πρέπει να περάσει σε ρόλο δευτεραγωνιστή. Αντιθέτω, ω προ την τεχνολογία, το δυναμικό καινοτομία, τι δημοκρατικέ μα παραδόσει και το σεβασμό για το κράτο δικαίου, αυτά ήταν παραδοσιακά οι αρχέ που έχουν ε, ε, τονώσει την επιτυχία τη Ευρώπη, το διεθνή ανταγωνισμό και ελπίζουμε αυτό να συνεχίσει να ισχύει. Παρ' όλα αυτά παραμένουν δύο προποθέσει. Μόνο μια Ευρωπαϊκή Ένωση που εσωτερικώ είναι ισχυρή θα μπορεί να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο διεθνώ. Μόνο μια Ευρωπαϊκή Ένωση που οικονομικώ είναι εξοπλισμένη θα μπορέσει να διατηρήσει την ε, δυναμικό τη χαρακτήρα. Εδώ, σε πολλέ περιπτώσει, έχουμε δει τι συμβολή μπορεί να προσφέρει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στι προσπάθειε τη Ευρωπαϊκή Ένωση να παραμείνει στην, ε, σε, πρωταγωνιστική θέση και στην, στον τομέα τη βιώσιμη ανάπτυξη εντάχει. Αντί να αντιδρούμε κύκλικα και να μειώνουμε τους όγκους ε, των επιχειρήσεων με τεράστιες προσπάθειες δανειοδότησης, για πρώτη φορά η τράπεζά μας είναι σε θέση με ένα τριετές πρόγραμμα να αντιμετωπίσει τις δραστηριότητες ε, χρηματοδότησης και δανειοδότησης, χάρη στην απόφαση των μετόχων να αυξήσουν το προκαταπευλημένο κεφάλαιο κατά 10 δις ευρώ. Αυτό το στηρίζει η πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία του Ευρωκοινοβουλίου και γι' αυτό σας είμαι ευγνώμων. Πέραν αυτού του νέου, της νέας ασπίδας θα δανείσουμε και 60 δις ευρώ πέραν και υπέρ των προηγουμένων στόχων. Αυτό θα φέρει το διεθνό, τον ετήσιο όγκο για το 2013-2015 στα 65 έως 70 δις ετησίως. Θα στηρίξουμε την οικονομία της γνώσης, τα προγράμματα για την οικοδόμηση υποδομών, την δράση για το κλίμα και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πέραν αυτών των επιπλέον κονδυλίων, αυτά θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά στα 27 και σύντομα 28 κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να στηρίξουμε την ανάπτυξη και τι ε, θέσει εργασία. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι θα αποχωρήσουμε από τον υπόλοιπο κόσμο. Αντιθέτω, εγώ θα ήμουν προσωπικά κατά τη τάση αυτή και το Ευρωκοινοβούλιο ελπίζω ότι σε αυτό θα είναι σύμμαχό μου. Και μάλιστα αυτή η Επιτροπή περισσότερο από κάθε άλλη. Εδώ και 50 χρόνια ο προπολογισμό ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τι εξωτερικέ πολιτικέ έχει συμπληρωθεί από τι μακροπρόθεσμε επενδύσει τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Με ε, επενδύσει σε τοπικό επίπεδο στι υποδομέ και στη δράση για το κλίμα. Από τα 52 δι ευρώ τη ΕΤΕ ε, το 2012, τα 7 κατευθύνθηκαν σε περιοχέ εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση και στην, στο πεδίο δράση τη ΕΤΕ, δηλαδή στην άμεση γειτονία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και την Ασία, τη Λατινική Αμερική και τι χώρε και μέσω των διεθνών μας συμφωνιών. Αυτό είναι ένα σημαντικό ε, ποσό σε σχέση με την εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το σχεδιασμό της. Έτσι, η νέα εντολή για δανειοδότηση σε εξωτερικέ δράσει ελπίζουμε θα στηριχθεί και από εσά και από τα κράτη-μέλη, χωρί να μειωθεί τα ερχόμενα χρόνια. Θα συνεχίσουμε να διευρύνουμε το 10% τη συνολική δανειοδοτική μα δύναμη στι χώρε εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζουμε ότι αυτό Ελπίζουμε ότι αυτό θα φέρει σημαντικά ωφέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρίε και κύριοι, όταν λέω 10% του όγκου δανειοδότηση, αυτό φαίνεται μικρό ποσό. Αλλά αν το συγκρίνετε με το τι συμβαίνει εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση και με άλλα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, θα αντιληφθείτε ότι η τράπεζά μα είναι τριπλάσια από την Παγκόσμια Τράπεζα σε δυναμικό. Και αν δείτε τι αριθμούς ε, αφιερώνουμε εμεί στην εξωτερική δανειοδότηση και το συγκρίνουμε με τις ε, πολυμερεί ε, τράπεζες ανάπτυξη. είμαστε οι μεγαλύτεροι μεταξύ τους. Το 10% λοιπόν μπορεί να σημαίνει πολλά διαφορετικά πράγματα. Ξεκινάμε από πολύ υψηλές βάσεις ούτω ή άλλως και μάλιστα συνοδεύεται η βάση αυτή από τον αριθμό 10. Στηρίζοντα την οικονομική ανάπτυξη παγκοσμίω, η ΕΤΕ συμβάλλει στο διεθνέ εμπόριο και δημιουργεί βάσει για τι ευρωπαϊκέ εξαγωγέ. Στηρίζοντα ε, ξέν, τι ξένε άμεσε επενδύσει, δημιουργούμε νέε αγορέ και επίση ένα ευρύ δίκτυο Ευρωπαίων πελατών παγκοσμίω, ώστε να ε, ενισχυθεί η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και ταυτόχρονα να έχουμε σοβαρά οικονομικά ωφέλη για τι ε, χώρε εταίρου. Επίση, με τι ε, διασυνδέσει των μεταφορέ και την ενέργεια με τι γειτονικέ χώρε, αυξάνουμε το επίπεδο ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επενδύοντα τι υποδομέ και την τεχνογνωσία για τι χώρε διεύρυνση, μπορούμε να προσφέρουμε και εκτιμένο και πρότυπα ευρωπαϊκά και σε αυτέ. Και με τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια και τι επενδύσει αυτό, πάλι διατηρούμε τον πρωταγωνιστικό μα ρόλο στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Κυρίε και σε έναν κόσμο που όλο ένα και περισσότερο είναι αλληλο, αλληλέν, αλληλεξαρτώμενος στο επίπεδο των κρατών μεταξύ τους. Η άμεση γειτονία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ιδιαίτερη σημασία για την ευημερία μας. Η ΕΤΕ δίνει μεγάλη σημασία λοιπόν στην οικονομική ολοκλήρωση και τη διαδικασία πρώτης προσχώρησης με την ευρύτερη πολιτική γειτονία και αυτό είναι μια από τις πρώτες μας προτεραιότητες εδώ και χρόνια. Η ΕΤΕ στηρίζει τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσπαθώντας να καταπολεμήσει τις περιφερειακές ανισότητες. Έχουμε σημαντικό ρόλο σε προηγούμενες διευρύνσεις. Να θυμίσω απλώς όταν η Ισπανία και η Πορτογαλία προσχώρησαν το 1986 και η χρηματοδότησή μας έχει πολύ, σημαντικές, ε, πολύ σημαντικά αποτελέσματα όπως φάνηκε και με τα 12 νέα μέλη το 2004 και το 2007. Το ίδιο τώρα ωφελούνται κράτες, ε, κράτη που είναι υποψήφια για την ε, προσχώρηση όπως η Κροατία. Το 2011 ξεκίνησε μια νέα πολιτική εποχή με την ε, πολιτική γειτονία προς τον Νότο. Οι χώρες ε, στο Νότο της Μεσογείου αξίζουν την στήριξη και την ενθάρρυνση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό πρέπει να ανοίξουμε τις αγορές μας και σε αυτούς. Ταυτόχρονα η δύσκολη κατάσταση στην ε, Αίγυπτο και τα τραγικά γεγονότα της Συρίας κάνουν τις περιοχές αυτές ακόμη πιο ευάλωτε και παθεί. Βέβαια το συμπέρασμα είναι ότι είναι τεράστιες επενδύσεις που χρειάζονται σε αυτή την περιοχή συνολικά. Τεράστιες προσπάθειες ε, αναδόμησης για να μπορέσουν να ξαναλειτουργήσουν οι χώρες αυτές είναι απαραίτητες. Όμω, για να κερδίσουμε πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών που βγήκαν στου δρόμου με τόσο θάρρο πριν από δύο χρόνια, πρέπει να του δείξουμε ότι υπάρχει και οικονομική προοπτική για αυτούς. Γι' αυτό έχουμε προσπαθήσει να δώσουμε απόκριση στι νέε κοινωνικέ, πολιτικέ και οικονομικέ πραγματικότητε. Από την Αραβική Άνοιξη και μετά έχουμε επαναλάβει την δέσμευσή μα στο νότο τη Μεσογείου σε πολλέ ευκαιρίε, μεταξύ άλλων τη ε, συνάντηση τη ε, δύναμη κρούση τη ε, Ευρωπαϊκή Ένωση Αιγύπτου τον περασμένο Νοέμβριο η μισή ε, δημοσιονομική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής στην όλη περιοχή ε, εκφράζεται σε δάνεια για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξη με κοινωνικές πτυχές ε, μέσω της πολυμερούς τράπεζας. 13 δις από το 2002, 1,7 δις πέρσι μόνο και 100 εκατομμύρια ευρώ για τεχνική στήριξη που λαμβάνει όλο ένα και μεγαλύτερη σημασία σε αυτό το πλαίσιο. Δεν υπάρχουν αρκετά κονδύλια στις περισσότερες περιπτώσεις και Ακριβώ αυτό που λείπει είναι η τεχνογνωσία. Με μεγάλη χαρά λοιπόν είμαι επικεφαλή μια τράπεζα που καλύπτει όχι μόνο το, τη διάσταση των τραπεζιτών, των οικονομολόγων, αλλά και επιστήμονες και φυσικούς και ε, εμπειρογνώμονες σε πολλούς διαφορετικούς τομείς. Είναι ζωτική σημασία αυτό. Είναι στατική σημασία σε όλη η περιοχή, στον νότο της Μεσογείου και ελπίζουμε ότι θα λάβει τη δέωσα προσοχή, όπως έγινε και προδιετίας, με όλη τη στήριξη την οικονομική, τη δημοσιονομική και την πολιτική που χρειάζεται για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματά τους. Ε, και εδώ λοιπόν με 900 εκατομμύρια ευρώ από το 2012 προς τους ανατολικούς εταίρους, ένα ρεκόρ και 1,1 δις ευρώ συμπληρώσαμε την τεχνική στήριξη που χρειαζόταν. Θα θέλαμε να διατηρήσουμε το ρυθμό αυτό για να μπορέσουμε να επιδιώξουμε του στόχου τη πολιτική γειτονία τη Ευρωπαϊκή Ένωση προ Ανατολά. Ε, Επίση, η εξωτερική δανειοδοτική μα εντολή θα μα ενισχύσει στην προσπάθεια αυτή. Είμαι βέβαιο ότι το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή σα θα σταθούν δίπλα μας για να βρούμε τη σωστή ισορροπία ε, στι διάφορε προπτικέ και προτεραιότητε των πολιτικών γειτονία. Η βάση για όλα αυτά, βέβαια, κυρίε και κύριοι, είναι η εξωτερική μα δανειοδοτική εντολή. Η εντολή που αφορά τον προορισμό και τον όγκο των επενδύσεων μα εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύντομα θα υποβάλει πρόταση για το διάστημα 2014-2020. Η νομοθετική διαδικασία θα πρέπει να προχωρήσει ταχαίω, διότι δεν υπάρχει χρόνο και χρειαζόμαστε νέα εντολή ω τον Ιούνιο του 2014 το αργότερο, εάν θέλουμε να αποφύγουμε διακοπή στι εξωτερικέ μα δραστηριότητε. Τουλάχιστον μια διακοπή στην υπογραφή των ε, επιπλέον δανείων. Γνωρίζουμε ήδη ότι το επόμενο πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο και με τα κονδύλια που θα προβλέπει για τον, από τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι πολύ περιορισμένο. Μεταξύ των και αυτών ο τίτλο 4. Έτσι, θα, θα καταστεί ο ρόλο μα ακόμη πιο σημαντικό από ό,τι ποτέ. Οι μηχανισμοί τη Ευρωπαϊκή Ένωση, συνδυάζοντα τι δωρεέ από τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλου είδου δάνεια από την ΕΤΕ και άλλε πολυμερεί ε, πηγέ, θα διδραματίσουν εδώ καθοριστικό ρόλο. Ελπίζουμε ότι θα παραμείνει πρωταγωνιστικό ρόλο τη ΕΤΕ στην πολιτική μόχλευση τη Ευρωπαϊκή Ένωση και στην προβολή και τον αντίκτυπο που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση εξωτερικώ. Είναι ο μεγαλύτερο δωρητή η Ευρωπαϊκή Ένωση και παρά τον κατακαιρματισμό ή την κατάτμιση τη ασυνέπεια τη χρηματοδότηση, αυτό εξακολουθεί να ισχύει. Και θα πρέπει να αυξηθεί βεβαίω εδώ η αποτελεσματικότητα τη χρηματοδότηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κάλυψη των εγγυήσεων Λοιπόν από πολιτικής άποψης και ε, από τα κράτη-μέλη των ε, δραστηριοτήτων της ΕΤΕ είναι πολύ σημαντική και το εργαλείο αυτό δεν επιφέρει άμεσο κόστος στον αναπροπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης Να θυμίσω ότι μόνο δύο φορές χρειάστηκε να ανακτήσουμε τέτοια ποσά. όπως ε, με τα 60 εκατομμύρια που ζητήθηκε να επιστραφούν ή 9,3 εκατομμύρια ευρώ που ανακτήθηκαν αναδρομικά. Μια περίπτωση επίσης της επικαιρότητα που είναι και πολύ καυτή ε, μας έχει φέρει σε 60 εκατομμύρια ευρώ περίπου σήμερα. Κυρίε και κύριοι, ήταν εντυπωσιακή η μεταμόρφωση τη ΕΤΕ την τελευταία δεκαετία. Είναι ακρογωνίω λήθο των πολιτικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση η χρηματοδότηση και για την δράση, για το κλίμα και τι ενέργειε και των μεταφορών και αυτά ε, διαρκώς εντείνονται. Έτσι ε, θα πρέπει να παραμείνουμε ένας ιδιαίτερος θεσμικό, ένα ιδιαίτερο θεσμικό όργανο που έχει κατεξοχήν δημοσιονομικό ρόλο μαζί με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λογοδοτούμε προς το ελεγκτικό συνέδριο, την Όλαφ, τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως εδώ με τους εκλεγμένους αντιπροσώπους της Ευρώπης όπου διαρκώς έχουμε εντατικό διάλογο. Δίνουμε μεγάλη έμφαση στη συνεργασία μας με την ΕΕ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους υπόλοιπους δημοσιονομικούς χρηματοπιστωτικούς μάλλον οργανισμούς και του διμερείς, τους των κρατών μελών. Γι' αυτό θέλουμε να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία και με το Ευρωκοινοβούλιο. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε συνέπεια με τον προγραμματισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για να προετοιμαστούμε για το ερχόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο μέχρι να ολοκληρωθεί. Θέλουμε η απέτηση για την ΕΤΕ να μεταφερθεί και προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να έχουμε μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση για τον κοινό εφαρμοστικό κανονισμό που θα διέπει τις δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός Ένωσης. Δεν θέλουμε να χάσουμε εδώ τη στήριξή σα και να μην ξεχνάμε ότι η ΕΤΕ είναι τράπεζα τη Ευρωπαϊκή Ένωση που ε, θεμελιώθηκε βάσει τη συνθήκη τη Ρώμη. Με ιδιαίτερε τεχνογνωσίε, με ιδιαίτερη προσοχή και ε, πεδίο δράση, το μόνο χρηματοδοτικό ίδρυμα που δεν στηρίζει απλώ τι ευρωπαϊκέ πολιτικέ όπω ορίζει η συνθήκη ή οι αποφάσει των θεσμικών οργάνων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και την εξωτερική τη δράση. Να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν πλήρω το δυναμικό τη. Ε, δεσμευόμαστε από τι αποφάσει των άλλων θεσμικών οργάνων και τι δικέ σα προφανώ και είμαστε το μόνο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που ανεξάρτητα και αποκλειστικώς μπορεί να καθορίσει τις, ε, την αποτελεσματική χρήση των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κονδύλια για τα οποία υπεύθυνοι είστε εσείς. Σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Σαλαφράγκα θα κάνει την πρώτη παρατήρηση. Ε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, καλώς ορίσατε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να σας πω ότι σε προηγούμενη μετασάρκωση στο Κοινοβούλιο διατέλεσα αντιπρόεδρος ε, του, της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος υπό τον ε, συνάδελφο και φίλο Πέτερινγκ κατέβαλα προσπάθειες ανέκαθεν έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να έχει δραστηριότητα και αιτήσια έκθεση μέσω της οποίας θα μπορούσε να έρχεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να εξηγεί τα πεπραγμένα και τις δραστηριότητες. Νομίζω αυτό είναι καλό ε, στο δημοκρατικό έλεγχο και χαίρομαι κύριε Πρόεδρε για την ανάλυση όσο και το όραμα που μας ε, παρουσιάσατε για τις δραστηριότητες της τράπεζας. Δεν περιορίζεται μόνο αυτό στον προορισμό σας για αναπτυξιακό εργαλείο των κρατών μελών, αλλά ε, έχετε να διαδραματίσετε και ένα ρόλο για την κρίση. Και μάλιστα όχι στραμμένη προς το εσωτερικό της Ένωσης, αλλά αντανακλά και ακτινοβολεί και η εικόνα της Ένωσης προς το εξωτερικό μέσα από τις δραστηριότητές σα Αναφέρετε τρία στοιχεία και είναι σημαντικά και τα ποσά κατά τα άλλα. που αφιερώνονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό τι δείχνει ότι είναι πάρα πολύ εύστοχη η δράση της τράπεζας του χέρι ε, της του τριπλού α και θα πρέπει να συνάδει πλήρως και σε πλήρη συνέχεια να, να βρίσκεται με τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην εξωτερική πολιτική από τον κανονικό της προπολογισμό. Στη συζήτηση για τις δημοσιονομικές προοπτικές βέβαια μειώνεται λόγω της κρίσης η χρηματοδότηση της Ένωσης, αλλά είναι γεγονός επίσης ότι σύμφωνα ε, με την πολιτική συμφωνία του Συμβουλίου Υπουργών και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 3,3% αυξάνεται η κατηγορία, ο τίτλος 4 του προϋπολογισμού μας. Εντάξει, δεν είναι και για κοδονοκρουσίες, αλλά εάν δούμε τι γίνεται σε άλλους τίτλους και σε άλλα κεφάλαια, υπάρχει κάποια αύξηση ε, έστω και στοιχειώδης. Θα ήθελα λίγο να σας ρωτήσω κύριε Πρόεδρε για το πώς κατανέμονται τα κονδύλια από τη χρηματοδότησή σας εκτός της Ένωσης σε τρία κεφάλαια ε, θεμελιώδη ή βασικά, τα οποία και εσείς αναφέρατε στην τοποθέτησή σας. Το προεταξιακό μέσο των κρατών που φιλοδοξούν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υποψήφιες χώρες σύμφωνα με την παρούσα εντολή 2013-2015. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερον, τα κονδύλια που δίνονται στην πολιτική γειτονία και στους δύο κλάδους και προς Ανατολάς αλλά και προς Νότον. Θα ήθελα να σας πω ότι είχα την ευκαιρία μαζί με άλλους συναδέλφους της Επιτροπής μας να συνοδεύσω την κυρία Άστον ε, στην Αίγυπτο, η Ορδανία και την Ισία όταν ξεκίνησα τη δράση τους η Task Force και επίσης ε, χαιρετήσαμε την παρουσία της τράπεζας και την υπογραφή σημαντικών συμβάσεων. Λοιπόν, τι προβλέπετε όχι μόνο για την παρούσα εντολή μέχρι το 2015 αλλά και για την επόμενη σε σχέση με τις δημοσιονομικές προοπτικές πάντα. Πιστεύετε ότι θα περιοριστείτε ε, στη σημερινή κατανομή. Τα δύο τρίτα πηγαίνουν στην νότια γειτονία και το ένα τρίτο στην ανατολική. Ή μήπω προτίθεστε να εισαγάγετε κάποιες τροποποιήσεις για να υπάρχει και αυτό το πνεύμα ισορροπίας το οποίο αναφέρατε και στην αρχική τοποθέτηση. Και ένα τελευταίο κύριε Πρόεδρε, Πρέπει να σας πω ότι εγώ είμαι πρόεδρος ε, στην ε, Ευρωλατινοαμερικανική Συνέλευση και στο Σαντιάγο της ε, Χιλής είχα την ευκαιρία να συμμετέχω σε μια σύνοδο κορυφής εκεί. Ξέρω ότι η τράπεζά σας πέραν της γειτονίας και πέραν των υποψηφίων κρατών έχετε πολύ σημαντική δράση στη χρηματοδότηση έργων στην Ασία και τη Λατινική Αμερική και θα ήθελα να μου πείτε ποιες είναι οι προβλέψεις σας και πώς ε, σκέφτεστε να κατανείμετε τους πόρους σε αυτές τις δύο περιοχές του κόσμου. Γιατί ακούμε κάποια ανησυχητικά νέα ότι θέλετε λέει να περιορίσετε τα χρήματα που δίνετε στη Λατινική Αμερική. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Ελπίζω να είναι συνεχής, διαρκής και μόνιμη στις εργασίες μας και όπως είπα και από την αρχή, χάρηκα πάρα πολύ για το όραμα που μας παρουσιάσατε, τη θεώρησή σας και την ανάγκη να συμπληρωθούν τα χρήματα ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις δικές σας δραστηριότητες στην εξωτερική δράση και αν μπορείτε να μας βοηθήσετε να έχουμε μια πιο συνεκτική, πιο ορατή και πιο αποτελεσματική εξωτερική πολιτική. Ε, είμαι βέβαιος ότι θα το κάνετε. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Γκόμες, ε, καλώς ήρθατε κυρία Χόγερ. Εκτιμώ ιδιαίτερο τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει και έχει αναλάβει η τραπεζά σα. όπως για παράδειγμα στη χώρα μου, κάτι που ήταν ε, εμφανέ στην Πορτογαλία. Όμως σήμερα αυτό δεν αναγνωρίζεται με τον ίδιο τρόπο. Δεν λέω ότι φταίτε εσεί. η προτεραιότητα της δημιουργίας θέσεων εργασίας δεν φαίνεται πια. Ούτε η τόνωση της ανάπτυξης. Δεν είναι ευθύνη μόνο της τράπεζας, είναι η όλη φιλοσοφία. Για να μην πω το θεολογικό δόγμα που διέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι πιστεύουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κρύβεται πίσω από τις πολιτικές λιτότητας. Από αυτή τη σκοπιά λοιπόν δεν βλέπουμε την τράπεζα ούτε κανένα θεσμικό όργανο της Ευρώπης να κάνει αυτά που είχε υποσχεθεί. Να προωθεί την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας, την απασχόληση. Να σας ρωτήσω όμως για την ανανέωση της εντολής σας και την εξωτερική μας δράση. Όπως είπατε και ο ίδιος, επηρεάζεται από τη σημερινή οικονομική κρίση της Ευρώπης. Και καθημερινά βλέπουμε ότι το μόνο δεν είναι μόνο η αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης που διακυβεύεται, αλλά και η αξιοπιστία μας. Είναι εδώ ο ρόλος που έχει να διαγραμματίσει λοιπόν η τράπεζα. Το είπατε κι εσείς. Πώς λαμβάνει αποφάσεις όμως η τράπεζα και πώς εντοπίζει τα προγράμματα που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν. Χρησιμοποιείτε κριτήρια που έχουν ήδη θεσπιστεί μέσω της πολιτικής γειτονίας λόγου χάρη. Πώς προσδιορίζεται το αν τα προγράμματα ε, αντιστοιχούν και καλύπτουν τις ανάγκες της αρχής more for more. Θα έπρεπε να υπάρχει ε, μεγαλύτερη συνεργασία με το Κοινοβούλιο, περισσότερη συντονισμένη συνεργασία όπως είπατε και εσείς και το υπονοήσατε. Και λέγοντας more for more, δηλαδή περισσότερες προσπάθειες για περισσότερα αποτελέσματα, και εσεί μπορείτε να επηρεάσετε εδώ. Πρέπει να καταλάβουμε ότι για να υπάρξει περισσότερο εκδημοκρατισμό στι γενικέ μα χώρε θα πρέπει να πετύχει ε, και η μεταρρύθμιση. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ των προτεραιοτήτων που θέτουμε, δηλαδή το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του σεβασμού του κράτου δικαίου, τη σωστή διακυβέρνηση, τη εταιρική διακυβέρνηση, τη καταπολέμηση τη διαφθορά και ούτω καθεξής. Καταλαβαίνω και σημειώνω αυτό που είπατε. Η τεχνική αρρωγή είναι σημαντική. Δεν είναι μόνο η οικονομική διάσταση σημαντική, αλλά και η τεχνογνωσία. Εσεί εδώ διαδραματίζετε σημαντικό ρόλο. Τα γνωρίζουμε τα στοιχεία αυτά. Όμω το ερώτημά μου είναι πώ το. Ε, να θυμίζετε αυτό. Πώ επιλέγετε τι θα χρηματοδοτήσετε. Για συγκεκριμένα προγράμματα και γενικώ. Επίσης τα γενικά αυτά κριτήρια που είναι ένας οδηγός καθορίζουν και το τι θα κάνετε για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών, την ε, ασφάλεια των ενέργεια, της ενέργειας, τις υποδομές μεταφορών. Οι υπόλοιπε προτεραιότητε τη διακυβέρνηση, λοιπόν, κατά πόσον λαμβάνονται υπόψη και πώ ενισχύουν τι δυνατότητε των ε, χωρών εταίρων να παίξουν το ρόλο που πρέπει στην παρακολούθηση υλοποίηση των προγραμμάτων και την οικονομική λογοδοσία των κυβερνήσεών τους. Η τράπεζά σας δίνει τη δυνατότητα στους ομολόγους των χωρών αυτών, στους υπευθύνους των χωρών αυτών να παίξουν έναν αντίστοιχο ρόλο ώστε να ελέγχονται τα προγράμματα και τα κονδύλια να πηγαίνουν εκεί που πρέπει μέσω των προγραμμάτων. Και επίσης τι γίνεται με την παιδεία, την εκπαίδευση. Τι θέση κατέχει στις προτεραιότητές σας. Και τέλος, κάτι που θα που μπορεί κανείς να πει ότι είναι αυτό που βαρύνει περισσότερο από όλα, είναι η Κίνα παγκοσμίω. Και βάσει των κριτηρίων του ΟΣΑ που δεν χρησιμοποιεί η Κίνα, έχει δικά της κριτήρια και για την ενέργεια και για τις πρωτασύλλες. Πάντως κάτι που έχουν σίγουρα οι Κινέζοι και όλοι οι συνομιλητές τους το τονίζουν είναι η ταχύτητα με την οποία λαμβάνουν αποφάσεις για τη χρηματοδότηση. Ενώ όλοι καταλογίζουν στην Ευρώπη ότι είναι πολύ αργή, πολύ γραφειοκρατική, οι διαδικασίε της χρονοβόρες. Εσείς πώς το αντιλαμβάνεστε αυτό στην τραπεζά σας. Ευχαριστώ. lass doch einfach η κυρία Μπράτνερ. Ευχαριστώ. Καλώ ήρθατε κύριε Χόγερ. Χαίρομαι που είστε μαζί μας σήμερα. Ήθελα να θέξω μόνο ένα θέμα. Αναφέρατε περιοχές που δεν είναι πολύ ειρηνικές, όπως ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλήσατε για την διεύρυνση των δραστηριοτήτων σας στην Λιβύη. Σε ποιο βαθμό το project αυτό και ο προγραμματισμός σας για την εφαρμογή και για το follow-up έχουν ε, εμπλέξει και την όλη ανάλυση της κατάστασης που επικρατεί, ε, γιατί ουσιαστικά μιλούμε και για μεταφορές και για φυσικούς πόρους, μιλούμε δηλαδή για τεράστια project. Αυξάνεται το δυναμικό ή μειώνεται το δυναμικό ε, αναταράξεων σε αυτές τις συγκεκριμένες χώρες και Ποιο αναλύει αυτά τα δεδομένα για σας και πώς επηρεάζουν αυτά τη δική σας εργασία. Μπορείτε να μας δώσετε παραδείγματα όπου μπορεί να αλλάξατε κάποιο project λόγω ακριβώς ε, των, συνεπειών που θα είχε, των συνεπειών που είχε η ανάλυση που κάνατε για την κατάσταση της χώρας. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, Μας παρουσιάσετε μια πολύ ωραία εικόνα για τα όσα κάνει η ΕΤΕ. Ε, γι' αυτό πληρώνεστε βεβαίως και αυτό δεν είναι κακό. Αλλά θα ήθελα να ρωτήσω κάποια συγκεκριμένα ερωτήματα. Υποστηρίζετε τους νικητές ή υποστηρίζετε κοινωνικά project που είναι ουσιαστικά οι χαμένοι ή υπάρχει ένα μείγμα και των δύο και πώς το ορίζετε. Με δεύτερον, τι οικονομικά ωφέλη θέλετε να πετύχετε με τα δάνεια που δίνετε και πώς τα αξιολογείτε. Τρίτον, ποιος σας συμβουλεύει. Έχετε ένα μεγάλο ας πούμε ε, ε, γραφείο με πολλούς ε, εμπειρογνώμονες ή χρησιμοποιείτε τον ιδιωτικό τομέα και ψάχνετε αρρωγή από παγκοσμίως για να επενδύσετε τα κονδυλιά σας. Και μια που λέτε ότι είσαστε υπόλογοι σε διάφορους σημαντικούς οργανισμούς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης και της Επιτροπής μας, Ποιος ε, βλέπει, ποιος παρακολουθεί τα δικά σας όρια και κρίνει αν αυτή η υπηρεσία αξίζει αυτά που λέμε ότι αξίζει ή μήπω τελικά επενδύοντας σε όλα αυτά τα project που δεν εγγυώνται οποιοδήποτε εισόδημα οικονομικό, πολιτικό ή κοινωνικό χάνουμε τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Ε, Ευχαριστώ. Έχω ένα ερώτημα να θέσω. Είναι παρόμοιο με αυτό που έθεσε η κυρία Γκόμες και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι. Κύριε Πρόεδρε, κατανοείτε κι εσείς ότι ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ως εκπρόσωπος ε, εσείς ε, του δικού σας ε, οργανισμού βεβαίως ε, πρέπει να σας αναφέρουμε τα, τις ανησυχίες που έχουμε για διάφορα project, για καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, για ε, περιορισμό της ελευθερίας του λόγου που υπάρχουν σε διάφορες χώρες. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πείτε πώς ακριβώς αξιολογείτε όλα αυτά τα στοιχεία όταν κάνετε το σχεδιασμό για τον δανειοδότηση από την τράπεζά σας. Προφανώς κάποιες, ε, άλλες, κάποιες πτυχές είναι πιο σοβαρές, κάποιες είναι λιγότερο σοβαρές. Αλλά για τους αρχηγούς πολλών ε, χωρών αυτό το εργαλείο είναι ιδιαίτερο σημαντικό και για μας βεβαίως είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο αυτό ειδικά όταν έχουμε τις, να αντιμετωπίσουμε τις σχέσεις αυτές ε, με αυτές τις χώρες. Μπορεί να ξέρετε να μην το γνωρίζετε ότι στην, στο Λονδίνο το θέμα των μπόνους των τραπεζιτών είναι τεράστιο ζήτημα και μάλιστα κάποια στιγμή το Κοινοβούλιο στην έκθεση Λάμπερτ ψήφισε για ένα όριο, ανώτατο όριο. Για τα μπόνους λοιπόν, εσείς στη δική σας τράπεζα δίνετε τεράστια μπόνους στο διοικητικό σας συμβούλιο ή έχετε, έχετε αγγλοσαξονική προσέγγιση, δηλαδή 5-10 φορές πάνω από τον μισθό τους ε, τον πόνους των τραπεζιτών σας ή έχετε, είναι απλώς ένας μισθός τον πόνους που παίρνουν. Μετά, το θέμα των πόρων για την Αίγυπτο ας πούμε και για την ειδική εντολή. Και επίσης ε, η δουλειά που έχετε κάνει σε σχέση με, την, ε, με τις ανατολικές χώρες και την εταιρική σχέση. Επιχειρησιακά Πώς ε, λειτουργείτε, πώς συνεργάζεστε με την ε, EBRD ε, και έχετε καλές σχέσεις για τη συγχρηματοδότηση τέτοιων project. Καταλήγετε στα ίδια συμπεράσματα ή υπάρχει και ένταση μεταξύ σας όταν σχεδιάζετε την χρηματοδότηση. Um, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω καλοπροαίρετα. Ίσως να μην καλύψω όμως όλα, να μην καταφέρω να τα καλύψω όλα. Εάν λοιπόν οι προσδοκίες σας δεν ικανοποιηθούν, θα σας ενημερώσω γραπτός. Ή μπορείτε να κάνετε και ερωτήσεις. Έχω πολλές απαντήσεις για, τα για την επόμενη μια μισή ώρα, οπότε Παρακαλώ για την υπομονή σα. Ο κ. Αλαφράγκα αναφέρθηκε στο βασικό ερώτημα, το κρίσιμο ερώτημα τη σημασία τη εξωτερική εντολή Είναι λογικό όταν ε, εκπροσωπώ την τράπεζα στο ΕΚΟΦΗΝ κάθε μήνα, υπάρχουν συνάδελφοι εκεί με διαφορετικέ προτεραιότητε. Θέλουν να ανακάμψει η ευρωπαϊκή οικονομία, να διευκολύνουν τι χώρε που αντιμετωπίζουν σοβαρέ πιέσει, Οι εξωτερικέ δράσει δεν είναι η πρώτη τους προτεραιότητα για τους περισσότερους υπουργούς οικονομικών. Αυτό δεν σημαίνει ότι το παραβλέπουν. Ξέρουν ότι θέλουμε μια πρωταγωνιστικό ρόλο για την Ευρώπη την ερχόμενη δεκαετία. Αλλά το θέμα είναι να θυμηθούμε εδώ πόσο τολμηρή ήταν η απόφαση όταν διπλασιάσαμε το, ε, ε, το κεφάλαιο της τράπεζας πέρσι, διότι μόνο τα 11 δις είχαν καταβληθεί ως τότε. Το διπλασιάσαμε το κεφάλαιο αυτό. Στις περισσότερες χώρες χρειάστηκαν κοινοβουλευτικές διαδικασίες με πολύ στενά όρια στον προπολογισμό τους εκείνο τον καιρό, με μεγάλες δημοσιονομικές πιέσεις. Ήταν επίτευγμα τον καιρό εκείνο. Φυσικά καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να επικεντρωθούν στην ευρωπαϊκή οικονομία. Το καταλαβαίνουμε όλοι, είναι κατανοητό. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να σεβαστεί τι υποχρεώσει τη πρώτα απ' όλα στη γειτονιά τη, στι γειτονικέ χώρε, σε αυτού που θέλουν να προσχωρήσουν. Αλλά είναι και στρατηγική σημασία το τι θέση θα δώσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προκύπτει και από τι διεθνεί μα συμφωνίε. Ο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ο πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Λέδη Άστον συνεχώς ταξιδεύουν στο εξωτερικό και έχουν ε, διαρκώ επιστρέφουν με ένα σωρό υποχρεώσει και συνεχώ το λογαριασμό τον πληρώνει κάποιο στο Λουξεμβούργο. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτή την εξωτερική εντολή και τη στήριξή σα. ο λόγο είναι 90 για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 10 εκτό. 5,5% για τις χώρες της προσχώρησης και τα υπόλοιπα για τις μοχλευμένες πολιτικές, για την ε, διοίκησή μας. Δεν μπορώ να αποθαρρύνω αυτούς που επικρίνουν. Περισσότερα χρειαζόμαστε. Να συνεχίσετε να επικρίνετε. Για τη Λατινική Αμερική τώρα. Είναι δύσκολα τα πράγματα εκεί. Αλλά είμαι αρκετά αισιόδοξο. Γιατί είναι από τις περιοχές όπου μπορούμε να είμαστε δραστηριοί. Όπω στι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, την ενεργειακή αποδοτικότητα, τι νέε ενεργειακέ πηγέ. Εκεί η συνεργασία με τη Λατινική Αμερική είναι εφικτή. Και υπάρχουν περιορισμοί, αλλά σκοπεύουμε να συνεχίσουμε τι προσπάθειε. Οι σχέσει μεταξύ η ισορροπία μεταξύ τη πολιτική γειτονία προ Ανατολά και προ τον Νότο είναι ευαίσθητη. Αλλά καθορίζεται και από το Συμβούλιο και από αυτή τη σκοπιά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμεί οι ίδιοι Λαμβάνομαι απλώς πολύ σοβαρά υπόψη τις αποφάσεις σας. Είναι κατανοητό για μένα. Ήταν έκπληξη η Αραβική Άνοιξη. Και η αναγνώριση σφαλμάτων των Ευρωπαίων από τους Ευρωπαίους ότι, που είχαν παραγνωρίσει το δυναμικό της Αραβικής Άνοιξης και το περιβάλλον που δημιουργείται στη Μεσόγειο πλέον αυτό δεν πρέπει να μας οδηγήσει σε λάθος συμπεράσματα για την πολιτική μας προσανατολές. Διότι τη δεκαετία του 90 ξεκινήσαμε μια πολιτική κατεύθυνση να ακολουθούμε και δεν έχουμε ακόμη πετύχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ίσως η κυρία Μπάρτον μετά να προσθέσει κάποια αριθμητικά στοιχεία γι' αυτό. Τώρα γι' αυτό το ερώτημα που έθεσε η κυρία Γκόμες. Όταν ταξιδεύει κανεί ε, στι χώρε τη Μεσογείου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Πορτογαλία συμπεριλαμβανομένη, βλέπει κανεί ότι εκεί οι άνθρωποι ξέρουν τι κάνετε. Διότι τα μεγαλύτερα προγράμματα οικοδόμηση υποδομών έχουν χρηματοδοτηθεί από την ΕΤΕ και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Προσπαθούμε να είμαστε ιδιαίτερα ενεργοί στην Πορτογαλία και η σχέση μα με τι πορτογαλικέ αρχέ είναι πολύ καλή. Καμιά φορά βέβαια έχει να αντιμετωπίσει κανεί γραφειοκρατικού κόμβου που προκύπτουν από τη Λισαβόνα ή τη Λουξεμβούργο ή άλλα σημεία και πρέπει να του λύσουμε. Αλλά τη στιγμή που οι μικρέ εταιρείε ζητούν πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για χρηματοδότηση, εκεί πρέπει να παρέμβουμε εμεί. Ή με γενικότερα δάνεια διακρατικά για την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πάντω, η έλλειψη πρόσβαση στη δανειοδότηση είναι μεγάλη απώλεια για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα για την εξωτερική μα πολιτική, ήδη έχουμε ειδικό σύμβουλο πλέον για τα θέματα αυτά. Και πραγματικά θα ήθελα να είχαμε στενότερη συνεργασία πολλές φορές και μαζί σας και με το Συμβούλιο και με την ΑΕΔ. Αυτή τη στιγμή όμως έχουμε ένα διεξοδικό κατάλογο προτεραιοτήτων ε, από κοινού με την ΕΕ και έχουμε καλέσει τους εκπροσώπους της ΥΠΑ της ε, εκπροσώπου να συμμετέχουν στις συζητήσεις μας. Στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζάς μας υπάρχει εκπρόσωπος της κυρίας Άστον που παρακολουθεί τις συνομιλίες. Παρακολουθούμε λοιπόν πάρα πολύ καλά το τι συμβαίνει με την εξωτερική πολιτική και τη... πώς σχεδιάζεται. Η διαδικασία Επιλογή τώρα. Είναι και ενδιαφέρουσα και πολύ ιδιαίτερη. Τα προγράμματα τα οποία μας υποβάλλονται για κρίση πρέπει να εμπίπτουν σε κάποια τις κατηγορίες που έχουμε ορίσει. Την ε, τεχνολογία της γνώσης, την ε, ενεργειακή αποδοτικότητα, την δημιουργία επιδομών. τι πολιτικέ που αφορούν τι μικρομεσαίε επιχειρήσει ε, με την ευρύτερη έννοια ή μεγαλύτερε υποδομέ. Οι τέσσερις αυτοί τομείς είναι περίπου 25% ο καθένας του συνολικού μας χαρτοφυλακίου. Η όλη διαδικασία μετά λαμβάνει υπόψη όχι μόνο την οικονομική διάσταση και τα οικονομικά κριτήρια που θα τα αναφέρω έπειτα, αλλά και το περιβάλλον εντό του οποίου όλα αυτά υλοποιούνται. Είμαστε τράπεζα της Ένωσης. Και η Ένωση αυτή είναι προϊόν των όσων συνέβησαν με τον διαφωτισμό. Λοιπόν, δεν μπορούμε να υπολοιπόμεθα των προσδοκιών των πολιτών μα σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτο δικαίου, αλλά να ξεχνάμε τι θέσει εργασία. Είναι πρωτιστή σημασία, λοιπόν, να κοιτάζουμε τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια, λόγω χάρη, που επικρατούν σε αυτό το περιβάλλον. Το ίδιο και την συμμόρφωση με τα πρότυπα και τη διαφάνεια. Το έθεσε η κυρία Μπράντον. Δεν μπορεί κάθε πρόγραμμα να επιλέγεται ούτε να υλοποιείται. Διότι δεν μπορούμε να θέτουμε να τα δικά μας ιδανικά, τις δικές μας αρχές επιλέγοντας ένα πρόγραμμα. Υπάρχουν προγράμματα που θα μπορούσα να δώσω ως παράδειγμα, αλλά υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις που απορρίψαμε προγράμματα προς επιλογή και αυτό θα θέλαμε να το διατηρήσουμε εμπιστευτικό. Υπάρχουν ακόμα και προσφυγές στο δικαστήριο για αυτά και εκκρεμούσε αποφάσεις. Η Κίνα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Βεβαίω υπάρχουν τα προβλήματα που μόλις αναφέρθηκαν. Αλλά ένα επιπλέον πρόβλημα είναι ότι οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ε, οι πρώτοι στόχοι της περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής, θα μπορούσαν να ενδυναμωθούν, θα μπορούσαν να προωθούνται μέσω τη συνεργασία με την Κίνα περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη μορφή συνεργασία. Οι ελάχιστε επενδύσει τη Κίνα στον τομέα τη καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών θα μπορούσαν να έχουν τεράστιο αντίκτυπο. Επιπλέον, αυτό που συμβαίνει στην Κίνα είναι ότι εκεί δεν είναι το πρόβλημα η έλλειψη χρημάτων. Έχει τεράστιο αποθεματικό η χώρα. Αυτό που συχνά λείπει είναι η τεχνογνωσία και το νομικό πλαίσιο για να οι δράσεις τους. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις διαφορών που κρίνονται αυτή τη στιγμή ε, στον ε, ΠΟΕ που θα μπορούσαν από περιβαλλοντική άποψης να στέκουν αλλά είναι διαφορές εμπορικές η Κίνα λοιπόν θα μπορούσε να είναι σημαντικό συνεργάτη και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον για μα. Αυτή τη σκοπιά δεν την ξεχνάμε. Αν, δεν έχουν, αν και δεν έχουν γίνει αρκετά ω προ αυτή την κατεύθυνση ακόμη. Η Κίνα επίση είναι κάποιο που παρακολουθεί τι κάνουν οι άλλοι και αποφασίζει αναλόγω. Η τράπεζα δεν δανείζει όμω κρατικά κονδύλια. Κρατικά κονδύλια έχουμε στην άκρη του κεφαλαίου μα, αλλά αυτή είναι η βάση μα για να δανειστούμε χρήματα. Εμεί βγαίνουμε στι αγορέ στις χρηματοπιστωτικές, στις, ε, ε, στις αγορές με 70-80 ε, δις ευρώ. Στις αγορές ομολόγων. Οι επενδυτές των αγορών αυτών πρέπει να μπορούν να μας εμπιστευτούν. Πρέπει να μπορούν να εμπιστευτούν τη δυναμικό της τραπεζάς μας. Και το 50% των χρημάτων που αποκομίζουμε από τις κεφαλογικές αγορές προέρχονται από μη ευρωπαϊκές πηγές. Αυτό έγινε τουλάχιστον πέρσι. Οι αγορές λοιπόν είναι για μας πολύ σημαντικές. Όχι μόνο των, ε, λόγω των οίκων ε, αξιολόγησης, διότι βλέπουμε πόσοι φορείς έχουν ε, υποβαθμιστεί, αλλά πρέπει να είναι πρόθυμοι οι επενδυτές να επενδύσουν σε μας. Έχουμε 500 δις, μισό τρεις στον συλλογισμό μας αλλά δυστυχώ και από τι δύο πλευρέ του συλλογισμού, όχι μόνο από τα έσοδα. Η εμπιστοσύνη λοιπόν των επενδυτών είναι διακύβευμα. Και βεβαίω θέλουμε να έχουμε παγκόσμια δυνατότητα. Η, η απονία λόγου χάρη, στι συζητήσει μα περί οικονομικών είναι κάτι που διαρκώ το ξεχνάμε. Είναι τεράστιο επενδυτή τη ΕΤΕ. Και οι Κινέζοι. Δεν πρέπει ούτε αυτά να τα ξεχνάμε. Ίσως θα ήθελες εσύ να απαντήσεις, ε, Τόμσεν, στην ε, ερώτηση της κυρίας Μπραντνερ και τα πιο συγκεκριμένα ζητήματα. Ίσως να μπορούσες να πεις κάτι γι' αυτό. Νομίζω ότι σχεδιάγραφησα μια ε, όντως καλή εικόνα της τράπεζας γενικώ, αλλά όντως είναι και ωραία η εικόνα. Είναι ένας ένα αξιόπιστο ίδρυμα με πολύ καλές επιδόσεις μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω. Αλλά ο στόχος μας δεν είναι να έχουμε τα μεγαλύτερα δυνατά κέρδη. Θέλουμε να τονώσουμε και τον ανταγωνισμό. Και αυτό φαίνεται από τα κέρδη που έχουμε, τις επιστροφές, τις εισρωές. Πέραν της κεφαλικής αύξησης όμως, και τη ενίσχυση τη κεφαλαιοκική μα βάση. τα κράτη-μέλη δεν έκαναν κάτι προ αυτήν την κατεύθυνση. Τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία συγκεντρώσαμε αρκετά κέρδη για να έχουμε ένα ευρύτατο πεδίο δραστηριοτήτων ακόμη. Για την ώρα πάντω, έχουμε πολύ γερέ βάσει. Δεν είχαμε απώλειες ως τώρα. Γενικώ ε, στον τραπεζικό κλάδο αυτή τη στιγμή πολλά δάνεια δεν αποδίδουν το τελευταίο διάστημα. Εμείς έχουμε ελάχιστες απώλειες σε ε, δεκαδικά ψηφία όμως θα μπορούσαν να μετρώνται αυτές οι απώλειες και είχαμε ένα κέρδος 2,7 ε, δις μόνο πέρσι. 70 μάλλον δις θα φτάσουμε από τα 50 προηγουμένως. Και βεβαίως έχουμε τριπλάσιο μέγεθος από την Παγκόσμια Τράπεζα. Με κάπως διαφορετικό πρόγραμμα βέβαια, ε, με αναπτυξιακό κυρίως πρόγραμμα εκείνη και με 10.000 εργαζομένους. Εμείς καταφέρνουμε τα τριπλάσια με 2.000 εργαζομένους. Ακριβώς γιατί έχουμε εξαιρετικά ειδικευμένου συμβουλου που καλέπτουν τι ανάγκε, αλλά πραγματικά η τεχνογνωσία μας είναι εντυπωσιακή. Βεβαίω, αυτό που μα απασχολεί είναι και το Συμβούλιο των Διευθυντών, το τι γίνεται δηλαδή με τα αφεντικά μα, το Συμβούλιο των Διευθυντών οι πρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών στις περισσότερες περιπτώσεις που συναντιόνται μια φορά το μήνα και κάθε πρόγραμμα, κάθε δάνειο περνάει από την κρίση τους. Τελικώς αυτοί που αποφασίζουν λοιπόν είναι τα κράτη-μέλη. Αλλά και η συνεργασία μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι στενότατη και πρέπει να είναι έτσι διότι μια από τις βασικές επιδιώξεις της τράπεζας είναι να βελτιωθεί η χρήση των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνδυάζοντας τα κονδύλια που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την δυνατότητα μόχλευσης στα δάνεια της ΕΤΕ. Γι' αυτό έχουμε στενότατη συνεργασία. Νομίζω παρακολουθούν στενά τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση το τι κάνουμε και το Κοινοβούλιο συμπεριλαμβάνεται βεβαίω σε αυτή τη διαδικασία. Ήμουν και στην Ολομέλεια, στο Στρασβούργο πολλέ φορέ και στη διαδικασία προπολογισμού συμμετέχω. Οπότε προφανώ έχουμε διαρκεί επαφέ με το Κοινοβούλιο. Ήδη θίξαμε τα, τα θέματα που αναφέρατε κι εσείς νομίζω, τα κριτήρια ρεσιμότητας λόγου χάρη. Τέλος πάντων για το τελευταίο σύνολο ερωτήσεων ε, για, το, για τα μπόνους των ε, τραπεζιτών και το τι γίνεται με τους μισθούς και τη συνεργασία μάλλον με την ε, Τράπεζα Ανάπτυξης και Έρευνας. Έχουμε πολύ καλή συνεργασία. Η συνεργασία μου προσωπικά με τον διευθυντή της τράπεζας αυτής είναι πολύ καλή. έχει σημαντικό ε, λιγότερο σημαντικό από εμάς η, BRD, αν και είναι πολύ στοχευμένη η δράση της, με μεγάλες επιτυχίες. Η αρχή πάντως είναι ότι η Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης δεν είναι ευρωπαϊκή. Οι Ρώσοι, οι Καζάκοι, οποιοδήποτε μη Ευρωπαίος συμμετέχει. Αυτό δείχνει πόσο τους ενδιαφέρει ούτως ή ε, η ανάπτυξη της Ευρώπης και για την Ευρώπη ξέρουμε τη σημασία της, της ανάπτυξης προς ΛΑΣ και προς τον Νότο όμως το ελεγκτικό συνέδριο, το δικαστήριο, το Ευρωκοινοβούλιο συμμετέχουν στη δική μας ε, δράση και ε, είναι διαφορετικά θεσμικά η διοργάνωσή μας. Τώρα για τα μπόνους τα όρια θεωρητικώς έχουν συζητηθεί με το Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά αυτά δημοσιεύτηκαν πριν λίγες και απέχουν πόρο από αυτά που έχετε ακούσει αλλού. Και για την ε, Επιτροπή Διαχείρισης και για εμένα τον ίδιο, να ξέρετε ότι το πόνου μου είναι μηδενικό. Όχι ότι δεν ταξίζω, αλλά πληρώνουμε βάσει των όσων ορίζουν οι συνθήκε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τίποτε περισσότερο. Ευχαριστούμε κύριε Χόγερ. Να ακούσουμε και την συνάδελφό σας, γιατί πρέπει να συνεχίσουμε. Να κλείσω κι εγώ, λέγοντας δύο πράγματα, για το πρώτο σημείο που θέσατε, για τον διαχωρισμό μεταξύ των περιφερειών. Δεν θα μπω στα της πολιτικής, αλλά είναι σημαντικό να γνωρίζετε τι μπορούμε να κάνουμε και σε ό,τι αφορά και την δυνατότητα απορρόφησης που έχουμε είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι έχουμε ε, φτάσει περίπου το 1 δις ευρώ πέρσι ε, δανεισμό προς Ανατολάς. Βεβαίω, αν αποφασιστεί να αυξηθεί αυτό θα μπορέσουμε να το κάνουμε. Ε, και μας ε, θέσατε ερωτήματα για το more for more και για το less for less. Νομίζω ότι η ευελιξία είναι αυτή που θα παίξει εδώ σημαντικό ρόλο σε όλη τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Τώρα, για τις πόλεμε περιοχές και για την διακυβέρνηση. Και τα δύο αυτά θέματα εμείς, ε, μας, εμάς μας συμβουλεύει η Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων και οι εμπειρογνώμονες στις διάφορες αντιπροσωπείας για το πού μπορούμε και πού δεν θα πρέπει να δανείσουμε. Αλλά σε ό,τι αφορά τα project έχουμε διάφορους μηχανισμούς, είτε είναι σε ό,τι αφορά την ευελιξία της περιοχής γιατί είναι σε εμπόλυμη κατάσταση, έχουμε συγκεκριμένες κατευθυντήρες γραμμές, έχουμε ειδικούς εμπειρογνώμονες που μελετούν το θέμα αυτό. Εγώ έχω έρθει σε επαφή με πολλές ΜΚΟ που ενδιαφέρονται για τέτοια project και μάλιστα πρόσφατα ε, ενσωματώσαμε και το θέμα της ευαισθησίας, της σύγκρουσης ή της σύραξης που υπάρχει στην περιοχή στα κριτήριά μας. Για τη διακυβέρνηση τώρα. Έχουμε, λαμβάνουμε κάποια τεχνική αρρωγή, δεν είμαστε σαν την Παγκόσμια Τράπεζα που έχει upstream μακροοικονομική τεχνική αρρωγή. Εμείς ε, έχουμε, παίρνουμε συμβουλές και για, τις, ε, για τα ενεργειακά project και τα λοιπά και έχουμε και πολύ αυστηρό ε, έλεγχο για θέματα ξεπλήματος μαυροκλήματος, απατών τα λοιπά Και για την συνεργασία μας με την EBRD. Πριν από λίγα χρόνια θα είχατε ακούσει ίσως διάφορες ε, ιστορίες για κακή συνεργασία μεταξύ μας, αλλά αυτό έχει ενισχυθεί και σε, στο ύψιστο πολιτικό επίπεδο, αλλά και στο πιο πρακτικό πολιτικό, ε, επίπεδο, γιατί έχουμε ε, μονάδες που μελετούν τις λεπτομέρειες αυτής της συνεργασίας και σε ό,τι αφορά την συγχρηματοδότηση και βεβαίως πάντα προσπαθούμε να εμβαθύνουμε τη συνεργασία μας. Νομίζω ότι τέθηκε και ένα ερώτημα για, τις, ε, για τα project της ε, ΕΤΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο. 88 δισεκατομμύρια ε, ευρώ δανείστηκε το Ηνωμένο Βασίλειο από το 99 μέχρι σήμερα για 1.200 project περίπου. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον πρόεδρο Χόγερ που ήταν σήμερα μαζί μας και βεβαίως προσβλέπουμε στις περαιτέρω συζητήσεις και συναντήσεις μαζί σας. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Γκουαλτιέρη και ο υποφαινόμενος σας υποβάλαμε μια πρόταση έκθεσης. Πρέπει να αλλάξει ο τίτλος. Συνεισηγητές πρέπει να γραφτεί. Όχι εισηγητές. Δεν φταίει η διοίκηση, η δική μας γραμματεία, γενικότερα η διοίκηση. Είναι δύσκολο λογικές διατυπώσεις να τις βάλουν στα χαρτιά εάν ε, δεν συνάδουν με το εδάφιο 4 του συνημένου άρθρου 5. Έχουμε δύο εισηγητές. Συν εισηγητές λέγονται αυτοί. Και δεν μπορεί να γράψει η διοίκηση συν αλλά γράφει τον έναν εισηγητή και τον άλλον συν γιατί είναι ένα υπόρθρακι που το έχουν εφεύρει οι ίδιοι, καταλάβατε. Äh, ε, και κάποια στιγμή σηκώνει στα χέρια ψηλά η δίκη του Κοινοβουλίου κάποια στιγμή αποκτά τέτοιε διαστάσει που δεν χρειάζεται πια του βουλευτέ για να εργάζεται και να απασχολείται. Äh, der und ich haben... Λοιπόν, ο συνάδελφος Γκαλτιέρη και εγώ σα κάναμε μια έκθεση, έλεγα, για την οποία και στην οποία ε, θα λάβει θέση και ο Πιέρεμο. Σας καλωσορίζω και ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και είστε στη διάθεσή μας να ανταλλάξουμε απόψεις. Θα σας πρότεινα υπό το φως της συζήτησης αυτής τις επόμενες ημέρες πριν το στείλουμε τη Δευτέρα το κείμενο για τροπολογίες να ε, βάλουμε στο έγγραφο την, ε, ε, τα αποτελέσματα μάλλον της συζήτησης. Πήραμε και μια επιστολή της Επιτροπής Νομικής, Νομικών Υποθέσεων. έχει διανεμηθεί Καλό θα ήταν. Αφορά τον κανονισμό υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων και μάλιστα είναι στην απόφαση αυτό με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καλό θα ήταν να συνυπολογιστούν αλλά αυτά και να ληφθούν υπόψη. για να αντανακλώνται και οι δικές του απόψεις στο κείμενο. Τώρα, πώς έχει κατάσταση. Η υπηρεσία εξωτερική δράση. Ε, σε μία διετία ε, από την ίδρυσή της έχει κάνει πρόοδους. Δεν είναι δύσκολο να ξεφυτρώσεις ξαφνικά από το μηδέν, από το έδαφος. Υπάρχουν ε, δυσκολίες, υπάρχουν ευαισθησίες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πάντα. Για ποιο λόγο πρέπει να παντρέψεις, να συγχωνεύσεις την πλευρά του Συμβουλίου με τις Επιτροπής. Έχουν αλλάξει και αρμοδιότητες έχουμε και τους διπλωμάτες των κρατών μελών που πρέπει να μπουν μέσα, Και τουλάχιστον 30% πρέπει να είναι, 60% τουλάχιστον κοινοτικοί υπάλληλοι. Ε, το καταλαβαίνουμε. οι, διπλωμάτες ε, των κρατών μελών ήθελαν να ε, πάρουν τα φιλέτα της διοίκησης ε, και ε, η χαμηλόβαθμοι να είναι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την Ευρωπαϊκή Διοίκηση. Εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν έγινε. Ε, θα πει και ο συνάδελφος κάτι, ο κύριος Γκουαλτιέρη. Εμείς δεν θέλουμε γενικά να επικρίνουμε και αόριστα. Κάνουμε προτάσεις από τους διάφορους τομείς πώς μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση. Προτάσεις λέγω στα διάφορα κεφάλαια. Γιατί δυνακότητα και αποτελεσματικότητα ε, τη διοίκηση χρειάζεται πιο αποτελεσματική δομή και λειτουργία. Θα πρέπει να θυμηθούμε και κάτι άλλο. Γι' αυτό έχει σημασία με τις προθέσεις των κρατών μελών, τις οποίες θέλω να σχολιάσω. Η υπηρεσία αυτή δεν αλλάζει τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κοινοτική πολιτική σε τελική ανάλυση είναι υπόθεση της, καθήκον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άλλα θέματα, ε, τα θέματα ασφαλείας και τα στρατιωτικά, εντάξει, γίνουν πιο πολύ προς την πλευρά του Συμβουλίου. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης είναι μία ε, προσπάθεια ε, που απορρέει από τον το εκπρόσωπο που έχει τριπλή ιδιότητα πλέον για να ε, καταλήξουμε σε μια συνεκτική πολιτική. Μια δεκαετία ε, ζωή έχει αυτή η έννοια από τη συντακτική συνέλευση. Τότε είχαμε υπουργό εξωτερικό, μα όχι υπουργό, επίτροπο εξωτερικό, είπα το εκπρόσωπο, που δεν είχε ούτε χρήματα ούτε διοίκηση ε, και μια εναλλασσόμενη προεδρία. και αυτές οι τρεις ε, τώρα ε, αποστολές έχουν συνενωθεί σε ένα πρόσωπο χωρίς να αλλάξουν όμως οι αρμοδιότητες του εκάστοτε θεσμικού οργάνου. Και γι' αυτό θα ήθελα να προειδοποιήσω παρακαλώ να μην χρησιμοποιείται ως πρόφαση η αποτελεσματική λειτουργία και ε, σιγά σιγά να αποδυναμώνεται και να κενώνεται η κοινοτική διάσταση και να εθνικοποιείται. Όπω προτείνουν διάφορε χώρε και πρωτοστατεί εκείνη που γνωρίζω εγώ καλύτερα. Δεν είναι κάτι το υβριδικό, ε, δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Μάλλον δεν καταλαβαίνουν ότι η υπηρεσία εξωτερική δράση είναι ένα υβρίδιο ε, συμβουλίου και επιτροπή. Τα κράτη-μέλη θέλουν να το βάλουν στο συμβούλιο. Η πολιτική γειτονία ίσω είναι το πιο εύγλωτο παράδειγμα και το πιο εξέχονο, αλλά όχι το μοναδικό και θέλουν και εκεί όλες οι διαπραγματεύσεις που έχουν να κάνουν με συμφωνίες σύνδεσης και εταιρική σχέσεις, όλες οι βασικές πολυμερείς ε, συνθήκες να πάνε στο Συμβούλιο και να ξεφύγουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με εκπλήση που δεν βάλαν και το εμπόριο ακόμα εδώ. Μα εδώ είναι παρεξήγηση. Γιατί λέγουν τα κράτη ότι καθίστε λέει να σκεφτείτε ποιος εκπροσωπεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την είπατε εκπρόσωπο. Λένε τα κράτη-μέλη. Ε, αυτή είναι η παρεξήγηση και καταλαβαίνουμε. Η ύπατη εκπρόσωπος είναι, ξέρετε, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βασικό πρόσωπο. Και θα πρέπει να αναλαμβάνει και τα καθήκοντά της ως αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το ρόλο της και μπορεί να επηρεάσει όσο και να καθοδηγεί τις εξελίξεις. Αυτή η ιδέα κρύβεται από πίσω. Ταυτόχρονα τη βλέπουμε. Η πολιτική και στρατιωτική διαχείριση των κρίσεων ε, θα πρέπει λέει να συνενωθούν και να πάνε στην εξωτερική υπηρεσία, στο Συμβούλιο. Υπάρχουν και εδώ μερικές πολιτικές ομάδες που λένε προσοχή να μην τα αναμειγνύουμε αυτά πάρα πολύ. Να μην πάρει το πάνω χέρι ο στρατός, α πούμε, η στρατιωτική διαχείριση των κρίσεων από την πολιτική. Το θέμα είναι που κατανέμονται αυτά, που εντάσσονται οι αρμοδιότητες. Και εδώ τώρα τι έχουμε. Προς μεγάλη μου έκπληξη, μετά από δυόμιση χρόνια που είναι σε ισχύ η συνθήκη τη Αβώνας, Έχουν αλλάξει δραματικά οι ε, εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χτες είδα την τελευταία εκδοχή αυτών των εγγράφων των κρατών μελών και έχω πραγματικά θορυβηθεί. Μπορώ να καταλάβω ότι, πώς να το πω, ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης έχει κάποιους συνεργούς ε, στο εσωτερικό τη κράτη-μέλη, στο πλευρό των κρατών μελών. Αυτό το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω ανθρώπινα, όχι θεσμικά. Και υπάρχει και κάτι ακόμα. Για τη μεταβατική περίοδο, αυτό με το 30 και το 60% στο διορισμό των, ευρωπαϊκών, των Ευρωπαίων πρέσβεων συγγνώμη, παίζουν ιδιαίτερο ρόλο τα κράτη-μέλη. Τώρα θέλουν να το κάνουν και για τους αντιπροέδρους των αντιπροσωπιών της ε, Ένωσης στο εξωτερικό και το καλύτερο θα ήταν να το αφήσουμε 100% στα χέρια τους. Τότε θα ήταν εντάξει η κατάσταση και σαφής. Επλην όμω δεν είναι αυτό το εγχείρημα, ξέρετε. Δεν είναι αυτό οργάνωση των κρατών μελών. Μετά από αυτή τη μεταβατική περίοδο που ολοκληρώθηκε και ε, πιστεύω από του χρόνου τα μέλη όλων των θεσμικών οργάνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης και με τους διαγωνισμούς που γίνονται μπορούν και εξωτερικοί να υποβάλουν υποψηφιότητα. Αλλάζει η κατάσταση λοιπόν ε, σε σχέση με τα όσα ε, ε, ίσχυαν στη μεταβατική περίοδο. Θα πρέπει να έχουν δικαίωμα πρόσληψης στελεχών. Όχι τα κράτη-μέλη. Η ίδια υπηρεσία να στελεχώνεται από μόνη της. Με κριτήρια, και ως κοινοβούλιο θα πρέπει να πούμε ότι χρειάζεται ένα πνεύμα ε, να δημιουργηθεί έτσι ένα πνεύμα που να του ανήκει στο ίδιο σώμα αυτό που λένε στα γαλλικά corps d'esprit esprit de corps και να μην είναι πάντα πεσπασμένοι οι υπάλληλοι των κρατών μελών αλλά θέλουν να, να δηλώσουν ότι θα παραμείνουν μόνιμα ε, διότι ε, υπάρχει και ένα θέμα αφοσίωσης και πίστης των υπαλλήλων. Ο κάθε υπάλληλο παραμένει πιστός σε εκείνον που ε, ευθυνέται για τη σταδιοδρομία του. Αυτό είναι ανθρώπινο και είναι κλασική επιρροή των κρατών μερών. Και σε παλαιότερες εκθέσεις θεωρούσα ότι θα πρέπει να είναι κοινή η εκπαίδευση των διπλωματών κοινοτική. Ήταν μια παλιά μας πρόταση και θέλαμε να τη ξαναφέρουμε. Ένα τμήμα, ένα μικρό τμήμα της εκπαίδευσης του διπλωματικού σώματος να ε, γίνεται μια κοινή εκπαίδευση Ευρωπαίων και εθνικών διπλωματών έτσι ώστε να έχουν ακριβώς αυτό το αίσθημα του ανήκει στο ίδιο σώμα, στο ίδιο διπλωματικό σώμα. Είναι σημαντικό αυτό. Και θα πρέπει να το πούμε τι λέει και η συνθήκη. Τα κράτη-μέλη είναι ε, κάτω των κοινωνικών στόχων, των στόχων. Ε, κυριαρχούν οι κοινωτικοί στόχοι ε, και οι στόχοι της συνθήκης. Το λέει η ίδια η συνθήκη αυτό και το ορίζει. Θα πρέπει να δημιουργηθούν λοιπόν οι απαραίτητε προϋποθέσεις. Ήθελα να κάνω αυτή την πολιτική εισαγωγή γιατί έχουμε πολλά σημεία και μεμονωμένα που πρέπει να λάβουμε υπόψη και μικρότερα ε, Απλώ θέλω να βάλω λίγο τα πράγματα στη θέση τους και να σας πω ποιες είναι οι πολιτικές και οι πολιτικοί συσχετισμοί. Το λόγο έχει τώρα ο συνάδελφος Γκολτιέρη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ, σχολιάζοντας τα όσα είπατε, ξεκινώ λέγοντας ότι όντως αναγνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης είναι μια θετική, ένα θετικό βήμα και στον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε να λειτουργεί και όπως παρουσιάζεται την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κόσμο με τις εξωτερικές μας σχέσεις. Ξέρουμε τι σημαντικά αποτελέσματα επετέξαν και ξέρουμε πόσο ήταν η πρόκληση μεγάλη ήταν δύσκολο πρώτα απ' όλα να ιδρυθεί και να δημιουργηθεί η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ακριβώς λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα που έχει η υπηρεσία αυτή. Διότι και ευρύ πεδίο τον έχει, από την κοινή πολιτική ασφάλειας μέχρι την, τον σχεδιασμό δημοσιονομικών εργαλείων, μέχρι το γεγονός ότι είναι διακριτόμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά στενά συνδεδεμένο. Με πολύ ε, δύσκολο έργο λοιπόν, αλλά με τεράστιο δυναμικό να γίνει ένα ισχυρό εργαλείο, ώστε με συνεπή τρόπο να ε, ενισχύσουμε την εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προφανώς όλες αυτές οι δυνατότητες δεν έχουν αξιοποιηθεί ακόμα πλήρως. Και έτσι, με την έκθεσή μας, προσπαθούμε να διατυπώσουμε προτάσεις για να επιτρέψουμε στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να αναλάβει πλήρως το ρόλο της. Έχουμε και κάποιες τεχνικές παρατηρήσεις και προτροπές, αλλά εδώ ήθελα να σταθώ και να υπογραμμίσω τις επιπτώσεις, το πολιτικό ε, περιεχόμενο των προτάσεων. Προτάσεις που θεωρώ λογικές όπως αυτές των deputies, όπως αυτές της απλοποίησεις της διαδικασίας ε, εντολών, το τι γίνεται με τον rating officer και τον managing director που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση, τι αρμοδιότητες πιστεύουμε ότι πρέπει να έχει, περιφερειακές περισσότερο, και να σταθώ σε δύο συγκεκριμένα σημεία που βρισκόνται στον πυρήνα νομίζω του όλου προβληματισμού του πώς θα αναλάβει πλήρως το ρόλο της και η υπηρεσία αυτή για να ενισχυθεί η εξωτερική δράση της Ένωσης. Οι σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρώτα απ' όλα, στι Βρυξέλλες και με τις αντιπροσωπείες. Οι δυνατότητε τη διπλής ιδιότητα τη ΕΠΑ εκπροσώπου αντιπροέδρου τη Επιτροπής δεν έχουν αξιοποιηθεί πλήρω. Ε, σημείο το οποίο αφορά όχι μόνο το ρόλο της ΕΠΑ εκπροσώπου, το πώς θα ασκεί τα καθήκοντά τη ανεμπόδιστα ω αντιπρόεδρος της Επιτροπής και συντονίστρια τη δράση των Επιτρόπων ω προς την εξωτερική πολιτική, αλλά ω και προς τον ίδιο τον τρόπο λειτουργία τη ΕΕΔ. Νομίζουμε ότι η υπηρεσία αυτή θα πρέπει να εξοπλιστεί καλύτερα, ώστε να μπορέσει και η υπατή εκπρόσωπος να αναλάβει πλήρως τα καθήκοντά της ως αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το άλλο σκέλο έχει να κάνει με τι αντιπροσωπείε. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Το έχουν πει και συνάδελφοι που είχαν τέτοιε εμπειρίε. Έχουν εργαστεί σε αντιπροσωπείε και συμφωνούν ότι αυτό που ορίζεται επισήμω από την απόφαση αρμοδιότητα των επικεφαλή, των πρόεδρων αντιπροσωπιών και του προσωπικού των αντιπροσωπιών, όλα αυτά για την ώρα δεν έχουν μεταφραστεί σε συγκεκριμένη ε, δυνατότητα να υπάρξει συντονισμός, να αποφευθούν επικαλύψεις, επαναλήψεις. Πρέπει να ακολουθήσουμε και στην πράξη τη συνολική αυτή προσέγγιση, κάτι που αντιπροσωπείς δεν το κάνουν ακόμη. Έπειτα υπάρχουν και κάποια άλλα ευαίσθητα ζητήματα. Ένα ερώτημα που θα πρέπει να το θέσουμε στους εαυτούς μας, αυτό του προπολογισμού. Ο δημοσιονομικός κανονισμός λοιπόν και το πώς κάποιες αρμοδιότητες θα ανατίθενται. Είναι ζητήματα περισσότερο τεχνικά βέβαια, αλλά πάντοτε υπάρχει και ένα παρασκήνιο πολιτικό, ε, ένα πολιτικό υπόβαθρο. Εκεί θέλουμε να εκφράσουμε την τοποθέτηση του Κοινοβουλίου. Το άλλο ευρύ θέμα αφορά το θέμα της διαχείρισης κρίσεων, το πώς αποκρινόμαστε σε καταστάσεις κρίσεων. Εδώ έχουν επιτευχθεί σημαντικά βήματα πρόοδου. Πέραν του κειμένου της απόφασης και των όσων ορίζει για την AR, η e, platform, η situation room, όλα αυτά ορίζουν την δυνατότητα δράσης και συντονισμού της AR e στο ε, τομέα της διαχείρισης κρίσεων που δεν έχουν να κάνουν τόσο με την ε, κοινή ασφάλεια και άμυνα για την οποία έχουμε θετική αποτίμηση ούτως ή άλλως. Οι εξελίξεις αυτές όμως ακόμη δεν έχουν οδηγήσει σε συνεπή ε, οργανική διάρθρωση στις δράσεις του κλάδου αυτού. Έτσι επιστρέφουμε σε μια παραδοσιακή θέση του Κοινοβουλίου, κλασική μάλλον, που την εκφράσαμε και στις ε, διαπραγματεύσεις. Δηλαδή, διαφορετικά μέσα διαχείρισης απόκρισης της ε, κρίση, όλες οι υποδομές που διαθέτουμε θα πρέπει να ενοποιηθούν σε μια δομή κοινή και κατάλληλη που να επιτρέπει συντονισμό αποτελεσματικό μεταξύ των υποδομών αυτών και των υπόλοιπων όπου και να εντοπίζονται γεωγραφικά και όλων των υπόλοιπων υπηρεσιών που κάποιες φορές πρέπει να συμμετέχουν στην διαχείριση κρίσιμων καταστάσεων. Αυτό είναι ένα πρώτο θέμα που δεν πρέπει να το συγχαίουμε με ένα άλλο. Έχει να κάνει με την κοινή πολιτική ασφαλείας και άμυνας και εδώ υπάρχουν ιδιαιτερότητε και ε, ανεξάρτητη εξέταση και από θεσμική άποψη με άλλη αλυσίδα εντολών που πρέπει να παραμείνει έτσι. Άρα να κάνουμε και εδώ βήματα πρόοδου. Αυτό επιθυμούμε και για να ενισχυθεί η δυνατότητα και ο στρατηγικός, το δυναμικό και ο στρατηγικός σχεδιασμός και μεταξύ του πολιτικού και του στατιωτικού σκέλους να υπάρχει αρμονία και να... παραλληλισμός στην αλυσίδα εντολών και στην επιχειρησιακή δράση. Θα πρέπει λοιπόν με την ενδέουσα σοβαρότητα, με την ε, επίγνωση των πραγματικών αναγκών στην πράξη, να αντιμετωπιστεί αυτή η έλλειψη ισορροπίας, παραλληλισμού. Δεν είναι ζήτημα τακτοποίησης νοικοκυριού απλού αυτό. Είναι θέμα του να αναλάβει πλήρως τις δυνατότητές της η εξωτερική δράση. Και ένα τρίτο πεδίο είναι το πολιτικό. Σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν το πρώτο σημείο. Συσχετισμός ΕΙΕΔ με άλλες υπηρεσίες και ιδίως των, με αυτές των κρατών μελών. Ένα τρίτο είναι αυτό που είπατε και εσείς Πρόεδρε και προσυπογράφω πλήρως. Αναφέρεται και στην εκθεσή μας. Χρήσιμη, μια χρήσιμη πρόταση της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων. Σε αυτά λοιπόν τα μεγαλύτερα ζητήματα και στην μετάφρασή τους σε πραγματική δράση. Εδώ θα θέλαμε τα σχόλια και της ΕΕΔ και του, των συναδέλφων. Ώστε να έχουμε μια συζήτηση επικοδομητική και να συνεισφέρει το Κοινοβούλιο στην δημιουργία μιας υπηρεσίας που να γίνει μια απόδειξη των επιτυχημένων προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά που ακόμη δεν έχει εξοπλίσει πλήρως τις δυνατότητές της. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κύριος Βημών, δεν θα πάρω πολύ χρόνο. Εγώ ήρθα να ακούσω περισσότερο εδώ παρά οτιδήποτε άλλο. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε και σας ευχαριστώ για την έκθεσή σας, το σχέδιο έκθεσης είναι πάρα πολύ χρήσιμο, είναι πολύτιμο θα έλεγα και άκρος ενδιαφέρον. Ε, από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης έχουμε αντίστοιχες ε, σκέψεις και εμείς και παρατηρήσεις και μας απασχολούν αυτό τον καιρό. Πρέπει να σας πω ότι Συμφωνώ πάρα πολύ με το επικοδομητικό και θετικό πνεύμα ε, που εσείς ο ίδιος υπογραμμίσατε κύριε Πρόεδρε και επίσης ε, ε, συμφωνώ απολύτως με τις αρχικές σας τοποθετήσεις που μας θύμισαν ότι σε θεσμικό επίπεδο θα πρέπει να τηρήσουμε τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες που απορρέουν από τη συνθήκη και με κανένα τρόπο να μην προσπαθήσουμε να τις υπονομεύσουμε. Σας διαβεβαιώ ότι και εγώ όπως και εσείς διάβασα το non-paper που κυκλοφόρησε από διάφορα κράτη-μέλη. Ε, δική τους θέση είναι αυτή, δεν είναι δική μας, ούτε της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Και για να είμαι ειλικρινή, δεν νομίζω ότι εμεί την εμπνεύσαμε με κανένα τρόπο. Έχουν δικέ του συνεδριάσεις και χαίρονται και πάρα πολύ. Είναι πολύ ικανοποιημένοι που προτείνουν τέτοια πράγματα. Κοιτάξτε, νομίζω ότι τρία είναι τα επίπεδα τα οποία πρέπει να μας απασχολήσουν. Ένα είναι το θεσμικό, δεν θα επανέλθω σε αυτό. Είπατε ε, όσα έπρεπε να υποθούν. Μετά υπάρχει το επίπεδο της όλης δομής και οργάνωσης και ε, οι δύο ε, το υπενηχθήκατε είναι ένα ζήτημα που πρέπει να μας απασχολήσει και να εργαστούμε και πάρα πολύ προσεκτικά, γιατί μπορεί να γίνει μεγάλη πρόοδος. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι αντιμετωπίζουμε, πώς να το πω, και κάποιες ιδιαιτερότητες και σε τεχνικό επίπεδο να λαμβάνουμε όλα αυτά υπόψη. Το παράδειγμα που είπε για την ΕΠΑ ο κύριος Γκαλτιέρη την ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας και άμυνας θα πρέπει να συντονίζεται καλύτερα και πιο αποτελεσματικά το εσωτερικό της υπηρεσίας και όλες οι υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με την διαχείριση των κρίσεων. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να γνωρίζουμε και να λαμβάνουμε υπόψη ότι οι μονάδες αυτές έχουν η κάθε μια τη δική τους εμπειρία, τη δική τους πραγματογνωμοσύνη, την οποία και αυτή θα πρέπει να τη σεβόμαστε. Θα πρέπει λοιπόν να βρεθεί ε, η σωστή ισορροπία ανάμεσα ε, στις διαφορετικές εμπειρίες και μετά στο πώς θα συγκεραστούν όλες αυτές μεταξύ τους. Ε, έχουμε κάνει μια πρόοδο ήδη, χρειάζεται και μεγαλύτερη. Αυτό είναι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, είναι ένα εργοτάξιο. Συνεχίζεται η προσπάθεια, έχουμε βεβαίως κάποιες επιτυχίες αλλά και πολλές αδυναμίες και θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε. Ίσως, αν μου επιτρέπετε, ε, μια φράση ακόμα για την εσωτερική μας ε, οργάνωση. Πριν από λίγες εβδομάδες ε, καλέσαμε τους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων Εξωτερικών και των 27 κρατών και ακούσαμε πολύ προσεκτικά αυτά που είχαν να μας πούν, σημειώσαμε και υιοθετήσαμε πολλά από τα σχόλια τους, τα επεξεργαζόμαστε αυτό τον καιρό. Αύριο Παρασκευή συνεδριάζει άτυπα το Υπουργείο ή το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών. Ε, θα έρθει και εσείς κύριε Πρόεδρε και χαιρόμαστε που θα συμμετέχετε κι εσείς. Το Και μετά... Θα προσπαθήσουμε να συντάξουμε μια έκθεση και τελικά ουσιαστικά θα είναι η έκθεση της υπάτης εκπροσώπου. Εκείνη θα κάνει τις προτάσεις της, ε, και τις ιδέες μετά από όλα αυτά. Βεβαίως θα σας στηρούμε ενήμερους και είμαι πρόθυμος να επανέλθουμε με τον David Σάλιβαν όποτε θέλετε για να σας ενημερώσουμε και να σας πούμε πώς προχωρεί η διαδικασία. Θα πρέπει ε, ε, να δούμε την πορεία και να προχωρήσουμε. Δύο τελευταία σχόλια για ορισμένα από τα όσα είπατε εσείς. Πρώτον, αυτό που ονομάσατε το ε, esprit de corps, ε, το αίσθημα του ανήκειν σε ένα συλλογικό σώμα. Θέλω να επιμείνω πάρα πολύ. Είναι πολύ δύσκολο αλλά και πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Ακριβώς πώς παντρεύεις τις δύο κουλτούρες, ε, τις δύο νοοτροπίες στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, ε, δηλαδή την εμπειρία και ό,τι κουβαλάει το προσωπικό του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ε, όλη την εμπειρία και το πλούτο που μεταφέρουν οι διπλωμάτες από τα κράτη-μέλη. Είναι δύο διακριτές ομάδες και αυτές θα πρέπει να συνεργαστούν καλύτερα, να συγκεραστούν καλύτερα για να δημιουργηθεί ένα ενιαίο σώμα. Αυτή είναι η προστιθέμενη αξία. Θα χρειαστεί κάποιο χρόνο όμως για να επιτευχθεί. Εμείς θέλουμε να αξιοποιήσουμε την εμπειρία όλων αυτών των πηγών που θα είναι κάτι διαφορετικό τελικά αυτό που θα δημιουργηθεί. Και όπως πολύ σωστά είπατε κύριε Πρόεδρε, τώρα μετά το 2013 που θα έχουν συμπληρωθεί δύο και τρία χρόνια λειτουργίας μας, θα έχουμε και άλλες πηγές τελέχωσης της υπηρεσίας και προσλήψεων, πολύ σημαντικές. Και όπως πολύ ωραία είπατε, λίγη τώρα κάπου η μεταβατική περίοδος και πάνω κάτω φτάνουμε στο στόχο του ενός τρίτου που είχαμε από τους ε, διπλωμάτες των κρατών μελών. Από εκεί και πέρα θα κανονίσουμε την πορεία μας. Θέλω να σας πω ότι όταν το συζητήσαμε αυτό με τα κράτη-μέλη, πολλά είπαν ότι θέλουν να επιστρέψουν οι διπλωμάτες τους που είχαν αποσπαστεί για μια τετραετία. Πολλοί από τους διπλωμάτες αυτούς πλέον έχουν εκπαιδευτεί και έχουν και μεγαλύτερη εμπειρία και πραγματονόμοσύνη στα ευρωπαϊκά θέματα και θέλει το διπλωματικό σώμα της χώρας τους να τους ε, ανακτήσει για να μπορέσουν να μεταδώσουν την εμπειρία τους και να τη μεταλαμβατεύσουν και σε άλλα στελέχη. Μακρηγόρησα πρόεδρε και σταματώ εδώ. Σας ευχαριστώ και πάλι που με καλέσατε. Ευχαριστώ. Εγώ μίλησα για Corps d'Esprit και εσύ μίλησες για Esprit de Corps. Αυτό είναι η διαφορά μεταξύ Γερμανών και Γάλλων. Thank you for reminding me, Das Wort hat der Ο κύριος Αλαφράγκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η δεύτερη συζήτηση για την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης μας δείχνει ξεκάθαρα Ποιε είναι οι προθέσεις του Κοινοβουλίου. Δηλαδή, βάσει της ε, εμπειρίας και των επιτευγμάτων, γιατί υπήρχαν και επιτεύγματα, και μόνο το γεγονός ότι δημιουργήθηκε αυτή η υπηρεσία εξωτερική δράση. Είναι πολύ μεγάλη κατάκτηση στην Ευρώπη. Είναι περίπλοκη η κατάσταση και δύσκολη και το εσωτερικό τη Ένωση. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μεγάλη επιτυχία. Τώρα, βάσει αυτή τη επιτυχία και από τα θετικά αυτά, αυτό που θέλουμε να κάνουμε να δούμε είναι με τι δεδομένε εμπειρίε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα και διδάγματα για να δούμε πώ μπορούμε να βελτιώσουμε αυτή την υπηρεσία. Θέλω να ακολουθήσω ότι η σειρά με την οποία μίλησε και ο πρόεδρος και ο κύριος Γκουαλτιέρη. Τρία πράγματα. Πρώτον, τα οργανωτικά, το δεύτερο είναι σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτον τα οικονομικά και τα θέματα του προσωπικού. Το οργανωτικό ζήτημα, Πρόεδρε. Νομίζω ότι μία από τις φόρμουλες που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε, όχι μοναδική βέβαια, είναι να εμπνευστεί κανείς από ε, ένα είδος ε, συμβούλιο, συμβούλιο εξωτερικών με την είπατε εκπρόσωπο, το Γενικό Γραμματέα ε, και κάποιους ειδικού εκπροσώπους. Το πρόεδρο της Πολιτικής Επιτροπής και Ασφαλείας και μαζί με το Γενικό Γραμματέα θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα κέντρο στρατηγικού σχεδιασμού που να εκτελεί αφενός τις ε, προτεραιότητες που έχει χαράξει το Πολιτικό Συμβούλιο, αλλά να κάνει και προτάσεις για να βελτιώνεται η δράση της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Πρόταση κάνω, μπορεί άλλος να κάνει πολύ περισσότερες. Αλλά για να ξέρουμε ποιες είναι αρμοδιότητες και ποια, ποια είναι η πολιτική δράση, αφενός ο πολιτικός προσανατολισμός και από την άλλη η διοικητική διαχείριση. Ο πρόεδρος δεν έχει ξεκαθαρίσει απολύτως ε, τη φύση του εγχειρήματο. Το είπε με μισόλογα. Ε, περί πρόκειται. Θα πρέπει να υπερασπίσουμε και να προασπίσουμε το κοινοτικό συμφέρον. Αυτό μας ενδιαφέρει. Δεν θέλουμε μια διακυβερνητική δομή ε, της υπηρεσίας. Κατανοώ ότι έχει μεικτή ε, φύση, αλλά αυτό που θα πρέπει να υπερασπίζεται είναι το κοινοτικό συμφέρον. Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου, όλες αυτές οι διευθύνσεις θα πρέπει να παραμείνουν ε, στην αρμοδιότητα και στην ευθύνη και στο πλαίσιο της ε, υπηρεσίας όπως τους αναλογεί. Η εκπρόσωπος μπορεί και θα έπρεπε ίσως να αναλαμβάνει περισσότερο τις ευθύνες της και ως αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Σώματος των Επιτρόπων και να το συζητάει και να συνεδριάζει μαζί τους. Τώρα, ε, ζούμε σε μια περίοδο κρίσης και θα πρέπει να αναζητήσουμε συμπληρωματικότητα με τα διπλωματικά σώματα των κρατών μελών. Παραδείγματα πολύ θετικά για τη χώρα μου έχει να κάνει με την Ιεμένη και τις κοινέ προξενικές αρχές. Επίσης υπάρχει και ο δημοσιονομικός ε, κανονισμός που λέγει ότι δεν χρειάζεται οπωσδήποτε να είναι ο επικεφαλής αντιπροσωπείας, μπορεί και ο αντιπρόεδρος. Ο κύριος Μπρόκ επίσης αναφέρθηκε και στα θέματα προσωπικού και στην ανάγκη να μην αποθαρρύνονται οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων πέρασε αυτή η μεταβατική περίοδος και άλλοι υπάλληλοι θα μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για την υπηρεσία αυτή από όλα θεσμικά όργανα, όχι μόνο από το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορεί να υπάρχει ένα σύνδεσμος ε, ή ένα σύμβουλος ε, που να είναι επιφορτισμένος για τις σχέσεις με το Κοινοβούλιο. Και Βεβαίω οι επικεφαλεί των αντιπροσωπιών θα πρέπει να επιλέγονται βάσει της προσήλωσής τους με το κοινοτικό συμφέρον, τη εμπειρία τους και τη διπλωματική εμπειρία βέβαια που έχουν οι εκπρόσωποι των κρατών μελών και μπορούν να βοηθήσουν όπως και βοηθούν άλλωστε και προσφέρουν ε, πολλά. Σε ό,τι αφορά το σύστημα επιλογή ή τα συστήματα κύριε Πρόεδρε για να είμαι ειλικρινή, η υπηρεσία εξωτερική δράση. Όταν επιλέγει επικεφαλής, νομίζω επέδειξε μεγάλη διαφάνεια. Εκπροσώπους επιζησίας εξωτερικής δράσης, ε, των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν ξέρω σε πόσα κράτη-μέλη αποφασίζεται έτσι ο διορισμός ενός, η, ε, η μετάθεση ενός πρέσβη. Εάν γίνεται με τόσο βαθιές διαδικασίες επιλογής. Πολλές φορές τα κράτη-μέλη γίνεται απλώς ψηφιακά και μόνο η μετάθεση. Εδώ νομίζω θα πρέπει να τους το αναγνωρίσουμε αυτό ότι ήταν προόδος. Όπως και άλλα όργανα τώρα ε, μπορούν να συμμετάσχουν στο προσωπικό, οι υπάλληλοι τους δηλαδή, ε, σίγουρα θα πρέπει να υπάρξει και μια επιλογή και να συμμετέχουν στα συμβούλια επιλογής και εκπρόσωποι των άλλων θεσμικών οργάνων. Επίσης, Πρόεδρε, πρέπει να αναζητήσουμε μία ισορροπία σε ό,τι αφορά... Τελειώνω, τελειώνω. Τελευταία σκέψη. Λέγω, μία ισορροπία σε ό,τι αφορά την εκπροσώπηση στα διοικητικά όργανα. Ε, τώρα, Γενικός Γραμματέας είναι διπλωμάτης από ένα κράτος μέλος. Είναι ο πιο κοινοτικό από του διπλωμάτες που θα μπορούσαμε να βρούμε. Οι δύο αναπληρωτέ είναι επίση διπλωμάτε από τα κράτη-μέλη. Αποτέλεσμα, να ομολογήσω κάτι. Στην πρώτη ε, συζήτηση άδικα επικρίναμε τον κύριο Σάλιβαν που διατέλεσε Γενικός Γραμματέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γενικός Διευθυντής Εμπορίου. Έχει πολύ μεγάλη εμπειρία και βοήθησε πάρα πολύ ε, να στηθεί αυτή η υπηρεσία. Λοιπόν, και το σκέλος το κοινοτικό θα πρέπει ε, ε ισότιμα και ισομερός να συμμετέχει, όχι μόνο τα διπλωματικά σώματα των κρατών μελών. Και δεν θα πρέπει να καταρακωθεί και το ηθικό των ε, Ευρωπαίων υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που τόσα χρόνια υπηρετούν πιστά και θέλουν να συμμετέχουν και αυτοί, όχι μόνο τα Υπουργεία Εξωτερικών των κρατών μελών. Η κυρία Γκόμες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για το σχέδιο έκθεσης. Θα το συζητήσουμε το γεγονός ότι ο Ρομπέρτο μαζί με εσάς το προετοιμάζει. Ήδη μας καθησυχάζει πολύ ότι έχετε κάνει πολύ καλή δουλειά. Θα ήθελα να πω ότι για μένα είναι ιδιαίτερο σημαντικό ως αποτέλεσμα όλης αυτής της αναθεώρησης και αυτό θα πρέπει να λέγεται ξεκάθαρα στο κείμενο η ύπατη εκπρόσωπος να ασκήσει το ρόλο που της έχει δοθεί από τη συνθήκη. Να είναι δηλαδή η συντονίστρια της Κομισιόν για τις εξωτερικές δράσεις. Να πάει δηλαδή και να φροντίσει ώστε οι, οι επίτροποι θα να σέβονται ε, την ε, πολιτική ε, καθοδήγηση που έχει η ίδια υποχρέωση να δίνει στους επιτρόπους σε ό,τι αφορά την, τις εξωτερικές δράσεις. Είτε είναι ανάπτυξη, είτε είναι εμπόριο, είτε είναι ενέργεια. Ό,τι και αν είναι. Αυτό νομίζω ότι είναι ζωτική σημασίας για να συμβάλλει και στη δημιουργία αυτού του αισθήματος ε, του ανήκειν που λέγαμε πιο πριν, το οποίο χρειάζεται βεβαίως. Αλλά πώς γίνεται να υπάρχει αυτό, αυτή η αίσθηση στις ε, υπηρεσίες αυτές, αν αυτό δεν υπάρχει στο ανώτερο δυνατό επίπεδο. Εμείς υποστηρίζουμε την ε, ύπατη εκπρόσωπο σε αυτό. Πρέπει να, να υπάρξει αυτό το αίσθημα για να υπάρξει και συνοχή στις πολιτικές μας και για να υπάρξει και αποτελεσματικότητα, επάρκεια ακόμη και σε θέματα χρηματοδότησης. Ξέρω ότι υπάρχει κεφάλαιο για τη χρηματοδότηση. Θα ήταν λοιπόν ενδιαφέρον να δούμε ποιο είναι το επίπεδο εκτέλεσης των μέσων χρηματοδότησης που έχουμε. Αυτό λοιπόν είναι ένα σημείο όπου αυτή η συνεργασία της ε, Υπηρεσίας Εξωτερικών Δράσεων με την Κομισιόν είναι ουσιώδης. Και δεν έχουμε σύμπραξη μέχρι στιγμή σε αυτών των δύο. Έχουμε αντίθεση μεταξύ τους. Πρέπει λοιπόν ε, οι ανώτεροι αξιωματούχοι να δώσουν πρώτοι το παράδειγμα. Μιλήσατε και για τους αναπληρωτές. Ακόμα και σε αυτούς τους καιρούς οικονομικών ε, ε, συμπληγάδων που βρισκόμαστε, ένας ε, αναπληρωτής είναι αρκετός. Βεβαίως η ύπαρξη αναπληρωτών είναι πολιτικό θέμα. Είναι πολιτικό θέμα. Και βεβαίως αυτό δεν, δεν αποκλείει το να είναι και πολύ εξειδικευμένος όπως ο εκπρόσωπος για τα ανθρώπινα δικαιώματα ή άλλα και να μπορούν να έρχονται όταν αυτό είναι απαραίτητο. Αλλά ένας αναπληρωτής με πολιτικό υπόβαθρο να μπορεί να εκπροσωπεί την είπατε εκπρόσωπο των αυτήν σε αποστολές στο εξωτερικό ή οπουδήποτε αλλού νομίζω ότι είναι σημαντικό να υπάρχει μια τέτοια θέση. Συμφωνάω με αυτό που είπε ο κύριος Σαλαφράγκα. Σε ότι πρέπει να δείξουν την πρωτοπορία σε ό,τι αφορά την ανάληψη και των ευθυνών των ίδιων των κρατών μελών από τα ίδια τα κράτη-μέλη. Μέσω των προξενικών ε, αντιπροσωπιών. Κάποια παραδείγματα είναι καλά, προφανώς έχουμε χάσει και κάποιες ευκαιρίες. Το Ιράκ, για παράδειγμα, έπρεπε για το Ιράκ να έχουμε κάνει μια κοινή προσπάθεια. προεβλέπετο, αλλά για οικονομικούς λόγους δεν ε, είχε αποτέλεσμα. Θα πρέπει όμως αυτό να, είναι, να αποτελέσει προτεραιότητα. Υπάρχουν και άλλες προτεραιότητες. Είχαμε προτείνει τη Βενγάζη. Μέσω του προξενείου εκεί. Ε, πρέπει να πούμε στην υπηρεσία ότι πρέπει να είναι διατεθειμένη και προετοιμασμένη ότι θα δουλεύει σε πολύ επικίνδυνα μέρη. Αν τώρα η θέση μας είναι ότι πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί με τους ε, κανόνες ασφαλείας, προφανώς δεν θα επιτύχουμε τίποτα και πουθενά. Αν οι διπλωματικές μας ε, αρχές πηγαίνουν μόνο σε πολύ ασφαλή και ειρηνικά μέρη, προφανώς δεν πρόκειται να γίνει δουλειά. Αυτό είναι ουσιώδες ζήτημα ναι, πρέπει να υπάρχει ισορροπία σε ό,τι αφορά τους ε, κινδύνους ασφαλείας, αλλά προφανώς θα υπάρχουν ε, κίνδυνοι. Το διπλωματικό επάγγελμα δεν είναι ασφαλές επάγγελμα. Είναι επικίνδυνο. Όσο επικίνδυνο είναι και το στρατιωτικό επάγγελμα και πολλές φορές και πιο επικίνδυνο. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουν και δεν θα πρέπει να αποτελεί αυτό περί, τροχοπέδι για τη δουλειά μας. Δεν μπορούμε να έχουμε πολύ αυστηρή πολιτική όπως έχουμε σήμερα και γι' αυτό δεν μπορούμε να είμαστε και αποτελεσματικοί. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνεισηγητές όπως σας λένε τώρα, η κυρία Γκόμες αναγνώρισε το έργο σας ε, δεν ξέρω βέβαια αν εμείς είμαστε τόσο ικανοποιημένοι μετά από όσα είπε η Άννα, αλλά στείλατε χτες το βράδυ αργά το κείμενο. Είχαμε το χρόνο να το μελετήσουμε, αλλά όχι να το συζητήσουμε μεταξύ μας, που σημαίνει ότι όλα όσα πω είναι προσωπικά σχόλια και ίσως οι συνάδελφοι να έχουν διαφορετική άποψη. Οπότε, σας το λέω για να το έχετε υπόψη σας. Σημερίζομαι την εκτίμησή σας και την ανέφεραν και οι προηγούμενοι συνάδελφοι ότι η δημιουργία της ΕΕΔ και η λειτουργία της ε, είναι από μόνο του ένα μεγάλο επίτευγμα. Έγινε εντός του χρονικού ορίου που είχε προταθεί, που για μένα ήταν πραγματικά θαύματο ότι συνέβη, και η λειτουργία είναι καλύτερη από όσο περιμέναμε. Παρόλο που προφανώς δεν έχουν ε, ε, πραγματοποιηθεί όλες οι προσδοκίες μας. Τα βασικά προβλήματα που τα περιμέναμε βέβαια και τα είχαμε προβλέψει κάποιοι από μας και οι υποφαινόμενοι ήταν ότι θα υπήρχαν προφανώς ε, διαχωρισμοί μεταξύ της, ε, των εθνικών ε, διπλωματικών σωμάτων και της, ε, και της ΑΕΔ. Ή θα, υπήρχε, θα υπήρχαν διαφορές μεταξύ της ΑΕΔ και της Κομισιόν. Αυτά τα είχαμε σκεφτεί, τα είχαμε προβλέψει. Ακούω τώρα ότι η σχέση μεταξύ ΑΕΔ και Γραμματείας του Συμβουλίου είναι πολύ ψυχρές, για να το πω έτσι, ευγενικά, ίσως να κάνω λάθος βέβαια, ίσως η πληροφόρησή μου να είναι λανθασμένη. Είναι ε, σημαντικό αυτό που λένε οι δύο συνσηγητές, ότι θα πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση σε ό,τι αφορά τις δομές της ε, Κομισιόν. Υποθέτω δηλαδή ότι αυτό σημαίνει ότι όταν επιμένουν ότι η ύπατη εκπρόσωπος, αντιπρόεδρος είναι αυτή που θα εκπροσωπεί όλους τους επιτρόπους που είναι υπεύθυνοι για θέματα που έχουν εξωτερικές πτυχές. Ότι δηλαδή αυτή θα κάνει αυτή τη δουλειά σε αντίθεση με το τι γίνεται τώρα που αυτό το αναλαμβάνει ο πρόεδρος της Κομισιόν. Ίσως βέβαια αυτό να περιπλέξει λίγο τα πράγματα. Επίσης πολύ διπλωματικά δεν λέτε τίποτα για τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και το κατά πόσο υπάρχει και εκεί κάποια διασύνδεση ή αν δεν υπάρχει. Όπως και να έχει εν πάση περιπτώσει το πράγμα, όταν, βλέ, όταν διαβάζουμε αυτό το non-paper του, το Υπουργείου Εξωτερικών, ε, βλέπουμε διαφορά απόψεων ανάμεσα σε αυτά που λένε αυτοί και σε αυτά που λέτε σωστά εσείς οι δύο συνεισηγητές. Είναι σαφές ότι το Υπουργείο Εξωτερικών αυτό το 30% των διπλωματών που προέρχεται από τις εθνικές αρχές ε, το θεωρούν ελάχιστο. Εμείς το θεωρούμε μέγιστο ποσοστό. 30% αν, έχει, αν το έχουμε φτάσει ε, σταματάμε. Αυτό είχαμε πει, οι ίδιοι το βλέπουν διαφορετικά. Θα δούμε τι θα γίνει και με την ψηφοφορία βέβαια. Αλλά όταν θα πούμε ότι τα κράτη-μέλη δεν έχουν ρόλο στην περαιτέρω επιλογή μελλοντικού προσωπικού, ε, προφανώς ε, τα Υπουργεία Εξωτερικών έχουν διαφορετική άποψη και θέλουν να συνεχίσουν να παίζουν το ρόλο που έχουν ή ακόμη και να τον αυξήσουν. Και επίσης υπάρχει και η πρόταση για την οποία δεν αναφέρεται κάτι μέσα στο κείμενο. Η πρόταση δηλαδή, η πολιτική γειτονία να ενταχθεί στο, στις αρμοδιότητες της ΙΕΔ ε, και το κατά πόσο εμείς το εγκρίνουμε αυτό ή όχι θα πρέπει να το δούμε. Δεν ξέρω τι κρύβεται πίσω από αυτό, κάτι θα πρέπει να κρύβεται πίσω από αυτή την πρόταση. Αλλά νομίζω ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα είναι αρκετά ικανοποιητικά. Πέραν αυτού, κύριοι συνεισηγητές, έχω δύο σχόλια για το ίδιο το κείμενο. Στο σχέδιο έκθεσης, στο J, στο G, μιλάτε για την επιχείρηση στο Μαλί. Και νομίζω ότι εκεί μπορούμε να πούμε πολλά. Είχαμε υποσχεθεί ότι θα το συζητήσουμε το θέμα αυτό και κυκλισμένων των θυρών. Δεν ε, ξέρω αν ε, είναι σωστό ή σοφό να ε, ωρεοποιούμε το πώς έχει πάει η κατάσταση στο Μαλί μέσα σε ένα εκτιμώντας μόνο, μέσα σε μια αιτιολογική σκέψη. Εγώ θα ήμουν λίγο πιο αυστηρή, αλλά εν πάση περιπτώσει θα τα δούμε. Και μετά έχουμε και το I, όπου γίνονται οι αναφορές στα EU Battle Groups και τα οποία δεν αναφέρονται πουθενά για, τις, για τους μάχημους σχηματισμούς. Υπάρχει και σχετική έκθεση που αναφέρει τους μάχημους σχηματισμούς, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο εδώ ταιριάζει αυτή η αναφορά. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για, την, για το σχέδιο έκθεση. Λίγα σχόλια για το σημείο 7 προτείνεται να συμπεριλάβουμε ε, και, την, ε, τα εργαλεία της εξωτερικής πολιτικής ε, στο, στην ΑΕΔ. Ε, νομίζω ότι είχαμε πει ότι το FBI θα μπει στις αρμοδιότητες του, της Ε.Ε αλλά χωρίς... Ε, αυτό όμως μονάχα, όχι οτιδήποτε άλλο το περιλαμβάνει. Δεν ξέρω, ίσως να είναι και η διατύπωση ε, τέτοια που μου δημιουργεί αυτή την αίσθηση. Μετά, σημείο 11. Υπηρεσίες ε, προξενικές. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε λίγο πιο ανοιχτοί σε ό,τι αφορά την συγχώνευση ε, προξενικών υπηρεσιών για να δημιουργηθούν ίσως ε, κάποια, κάποια pools, κάποιες ε, ομαδικές, ομάδες τέτοιων υπηρεσιών. Τα κράτη-μέλη ούτως ή άλλως στέλνουν πόρους στην υπηρεσία εξωτερικών δράσεων. Αν θέλουμε να δημιουργήσουμε τέτοιες ομάδες εντός των αντιπροσωπιών, αλλά χωρίς επιπλέον προσωπικό, δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό, σωστό αυτό που προτείνουμε. Μετά, στο σημείο 16. Είναι σημαντικό να υπάρχει το crisis response, η ανταπόκριση της κρίσης, γιατί βέβαια και η διαχείριση της κρίσης είναι ίσως κάτι παρόμοιο, αλλά παρόλα αυτά δεν είναι απολύτως ταυτισμένα. Είναι σημαντικό λοιπόν να υπάρχουν και τα δύο και ίσως καλό θα, πρέπει, καλό θα είναι να ορίσουμε τι σημαίνει το crisis response. Και στο 17 είναι πολύ καλή η διατύπωση της παραγράφου αυτής. Σε σχέση με αυτό που είπε και ο κύριος Βημό, ε, μπορεί ε, να, συγχωνεύσει κανείς ε, την εμπειρογνωμοσύνη. Το ποιος αποφασίζει δεν πρέπει να συγχαίουμε. Οπότε πρέπει να ξέρουμε τι μπορούμε να συνδυάσουμε και τι όχι. Είναι σημαντικό να, να συγχωνεύεται και να συνδυάζεται η εμπειρογνωμοσύνη από το CMPD και το CPCC. Είναι σημαντικά κέντρα. Αλλά το θέμα δεν είναι η εμπειρογνωμοσύνη και, και ο συνδυασμό τη. Είναι σημαντικό να μην ε, συγχέονται όμως ε, ε, οι, υπεύθυνοι. Και μετά στο σημείο 35 λέτε για καλύτερη ισορροπία φύλου και γεωγραφική ισορροπία. Στη σελίδα 2 ο κύριος Λένε λέει ότι στο εκτιμώντας 15 του κανονισμού η ύπατη εκπρόσωπος ε, έπρεπε να αναλάβει μέτρα ώστε να προωθηθούν οι ε, ίσες ευκαιρίες. Ε, αυτό δεν αναφέρεται ακόμα. Οπότε ίσως θα πρέπει να ρωτήσουμε τι έχει γίνει ως προς αυτό μέχρι τώρα. Και αυτό για τη Διπλωματική Ακαδημία που είπατε κύριε Μπροκ, στη δική μας την απόφαση υπήρχε μια παρόμοια αναφορά όπου μιλούμε για ένα, μια κοινή, κοινές δραστηριότητες ε, κατάρτισης, εκπαίδευσης, καθώς επίσης και αυτό το Esprit de Corps που αναφέρεται. Ακόμη δεν έχει γίνει κάτι ως προς αυτό. Αυτά από μένα και ευχαριστώ. Χωρίς μικρόφωνο, πρόεδρο. Um, Ο κύριο Στάνοκ, ευχαριστώ Πρόεδρε, αλλά εδώ σταματάει η διερμηνία, διότι ολοκληρώνει το ωράριο του η διερμηνία